Καλό απόγευμα σε όλους. Ελπίζω όλοι να ε, περάσατε καλά το μεσημεριανό διάλειμμα. Εγώ καλά το πέρασα και σας καλωσορίζω όλους καθώς ε, και όλους όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Δημόσια Κρόαση για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας με βάση όλες τις αναφορές που έχουμε ε, λάβει. Και χαίρομαι πολύ που σήμερα οργανώνει η Επιτροπή μας ε, αυτήν την εκδήλωση, διότι ελπίζω ότι θα απαντήσει έτσι σε πολλά ερωτήματα που έχουμε όλοι μας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάποιες πρακτικές πληροφορίες παρέχεται διερμηνία στις 24 επίσημες γλώσσες με κάποιες ε, εξαιρέσεις, τα εστονικά, τα φιλανδικά, τα λιθουανικά, πορτογαλικά, σλοβένικα, τσέχικα και κροατικά. Κατά τα άλλα, έχουμε διερμηνία σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Επίσης, παρακαλώ να γνωρίζετε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η ακρόαση αυτή και θα καταγραφούν όλες οι παρεμβάσεις ε, των ε, ομιλητών. Ε, αυτά ήταν τα πρακτικά ζητήματα. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην ακρόαση που θα δώσει την ευκαιρία στους ευρωβουλευτές, τους ομιλητές και το κοινό, όλους τους παράγοντες να σκεφτούν ε, τους διάφορους πολύπλοκους ε, τύπους ε, εργασίας και να βγάλουν άκρη με τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που υπάρχουν. Από την έναρξη της θητείας μας το 2014 η Επιτροπή μας έχει λάβει όλο ένα αυξανόμενο αριθμό αναφορών με ανησυχίες ε, εργαζομένων ε, με προσωρινή απασχόληση ή με επισφαλή θέση εργασίας. Ε, και οι αναφορές αυτές προέρχονται και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Πολύ... έχουν αναφέρει ότι για ίδια ή παρόμοια καθήκοντα λαμβάνουν διαφορετική αμοιβή και δεν καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας. Άλλοι ανησυχούν σχετικά με το γεγονός ότι το είδος τέτοιων συμβάσεων έχει γίνει κανόνας και τελικά αντικαθιστά πιο παραδοσιακές μορφές ε, μονίμων συμβάσεων. Και έτσι τώρα αυτές οι μορφές εργασίας ε, μετατρέπονται σε ε, προσωρινές θέσεις εργασίας. Θα ακούσουμε ε, λοιπόν σήμερα τους ομιλητές μας. Έχουμε την μελέτη για τις, προσ... για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η μελέτη έχει εκπονηθεί από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ κατόπιν εντολής της Επιτροπής μας και εξετάζει τη φύση και ε, την έκταση της ε, επισφάλειας ε, στην απασχόληση στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας περί απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται στις άτυπες μορφές απασχόλησης και τη δικαιοχρησία. Η ακρόαση θα ε, χωριστεί σε δύο τμήματα. Καταρχάς θα ασχοληθούμε με τις ε, θέσεις απασχόλησης ε, στην Ευρώπη το 2017 με ομιλητές από διάφορα πανεπιστημιακά κέντρα και ομάδες προβληματισμού και εκπροσωπούν διάφορες χώρες και διάφορες προοπτικές. Επίσης, μεταξύ των ομιλητών στο πρώτο τμήμα έχουμε έναν συνάδελφό μας, Ευρωβουλευτή από την Κύπρο, τον κύριο Σιλικιώτη από την Επιτροπή απασχόληση. Ε, χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Ε, και το δεύτερο τμήμα ε, επικεντρώνεται στο νομικό και κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο των επισφαλών και προσωρινών μορφών απασχόλησης. Κατά το τμήμα αυτό της ακρόασης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργοδοτών και αναφερόντων θα πάρουν το λόγο. Θα ε, έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μιλήσουν για ε, τις ε, συνθήκες εργασίας, την ευελιξία στις ώρες εργασίας και την ασφάλιση για τους εργαζομένους. Είμαι βέβαιη ότι αυτή η ακρόαση θα αποτελέσει πολύ καλή ευκαιρία για τα μέλη της Επιτροπής μας και τους προσκεκλημένους μας να προβληματιστούν πάνω στο ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα των συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Καταρχάς ε, έχω τη χαρά να δώσω το λόγο στην Αριστεία Κουκιαδάκη, ε, καθηγήτρια εργασιακού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μάνσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Ιωάννη Κατσαρούμπα. Και οι δυο σας ε, μένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εσείς είσαστε καθηγητής Εργασιακού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Θα μας παρουσιάσετε την ε, μελέτη του θεματικού τμήματος ε, ΓΑΜΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που μόλις ανέφερα. Δίνω το λόγο και στους δυο σας. Να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ομιλία. Πέντε λεπτά περίπου έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Um, uh, Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή που μας επιτρέπει, μας επέτρεψε να ε, εκπονήσουμε και να παρουσιάσουμε σήμερα αυτή την ε, μελέτη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την διοικητική ομάδα της Επιτροπής που μας ε, υποστήριξε στην προσπάθειά μας. Ε, τα θέματα σχετικά με τη, τα ε, συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ε, και την επισφαλή εργασία καθώς επίσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων άρχισαν να απασχολούν πολύ περισσότερο ε, την κοινή γνώμη με, την οικονομική κρίση. Η επισφάλεια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Ο, ο όρος άρχισε να αναφέρεται ακόμα και σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πιο, το πιο πρόσφατο αλλά και πιο σημαντικό παράδειγμα αφορά την ανακήρυξη του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, που έλαβε η χώρα στην περασμένη εβδομάδα στο Κέτεμπορκ. Στις, ε, ε, αυτό που προσπαθήσαμε είναι να εντοπίσουμε ε, με ένα σύνολο από γενικές ιδέες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις εξελίξεις και τις ε, συνέπειες τους ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, τα δικαιώματα και την επισφάλεια. Το πιο σημαντικό πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι πιστεύουμε πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Και αυτή η αλλαγή ε, έθεσε σε κίνηση και μια ε, διαδικασία ε, μετακίνησης των κινδύνων από μια σειρά οντοτήτων που είναι ο εργοδότης συνήθως αλλά και το κράτος στον εργαζόμενο. Με αυτόν τον τρόπο κατακαιρματίζεται η αγορά εργασίας και δημιουργούνται συνθήκες επισφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές τις οποίες εξετάσαμε στην έκθεσή μας, ε, φαίνεται αυτή η διαδικασία μεταφοράς, μεταβίβασης, ε, με αύξηση των, των διαφόρων άτυπων μορφών απασχόλησης όπως συμβάσεις ε, μηδενικού χρόνου κλπ. Ένα δεύτερο παράδειγμα μετακίνηση του κινδύνου αφορά την, τον κατακαιρματισμό των εργαζομένων, των εργαδοτών μέσω των δικτύων ε, franchise, ε, δικαιοχρησίας δηλαδή, ε, υπεργολαβιών κλπ. Αυτή η διαδικασία ε, μετακίνησης των κινδύνων ε, απαιτεί από μας να αναλύσουμε την επισφαλή εργασία ε, και να την, αντιμετωπίσουμε, να την αντιμετωπίσουμε ως ένα συνεχώς μετακινούμενο στόχο. Η επισφάλεια είναι ένα φαινόμενο που έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις και εξαρτάται και από πολλούς αλληλοεπιδρόντες και αλληλοεξαρτούμενους παράγοντες. Οπότε για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Στην έκθεση λέμε ότι το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε και θα έπρεπε να ερμηνεύεται ως ε, υποστηρίζον μιας ε, ε, αντιμετώπισης υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων εναντίον της επισφάλειας και υπέρ της προστασίας των εργαζομένων έναντι αυτής της επισφάλειας. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις και επί τη βάση των αναφορών που λάβαμε από την Επιτροπή, τι κάναμε. Δημιουργήσαμε ένα αναλυτικό, χρησιμοποίησαμε ένα αναλυτικό πλαίσιο που έχει χρησιμοποιήσει και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο ΑΕΛΟ, ε, που λαμβάνει υπόψη και τι αλλαγέ στην δομή τη οικονομίας και την υπάρχουσα νομοθεσία. Οπότε εντοπίσαμε τις διάφορες ε, διαστάσεις ε, κενών που υπάρχουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την προστασία της εργασίας. Ως ε, αποτέλεσμα του ότι ορισμένοι, ορισμένα άτομα δεν κατηγοριοποιούνται, δεν ταξινομούνται ως εργαζόμενοι, οπότε δεν μπορούν να απολαμβάνουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Δεύτερο κενό στην προστασία των εργαζομένων είναι το κενό στην αντιπροσώπευση. Αυτό έχει σχέση με καταστάσεις όπου ε, οι εργαζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση σε όργανα τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν τη φωνή τους, για παράδειγμα συνδικάτα ή, άλλα. Άλλες μορφές δημοκρατικής εκπροσώπησης. Τρίτο και κενό στην προστασία έχει σχέση με την εφαρμογή. Διαφορές στου τρόπου εφαρμογή τη νομοθεσία μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να μην γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα, τις συμβάσεις μηδενικού, μηδενικών ορών εργασίας. Αλλά μπορεί να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά να μην θέλουν να φοβούνται να τα ασκήσουν. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την ταξινόμηση την οποία έχει αναπτύξει ο ILO και άλλοι ερευνητέ για να διαπιστώσουμε πώς αυτά τα κένα, αυτές οι αδυναμίες ε, εμφανίζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξαμε το πρωτογενέ δίκτυο, ε, δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το δευτερογενέ δίκτυο, δίκαιο συγγνώμη, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώ η νομοθεσία των κρατών μελών αντιμετωπίζει αυτά τα κενά. Οπότε, ας εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε ε, ατομική διάσταση της ε, επισφάλειας. Έχει σχέση με τη χρήση αλλά και την κατάχρηση μη τυπικών μορφών εργασίας. Για παράδειγμα, συμβόλαια μηδενικών όρων εργασίας στο Ηνωμένο ε, συμβόλαια ε, ελαστικών συμβάσεων στο Βέλγιο ή και ε, συμβόλαια συμβάσεις περιορισμένου χρόνου στον κρατικό τομέα σε άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό το εξής. Είναι δυνατόν να εντοπίσουμε συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στην επισφάλεια και ε, ορισμένους νομικούς ή και μη νομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επισφάλεια. Μεταξύ αυτών το πρόβλημα της ε, πρόσβασης στα εργασιακά δικαιώματα, για παράδειγμα στην περίπτωση των συμβάσεων μηδενικού χρόνου εργασίας. Πρόκειται για κενά που υπάρχουν στα ατομικά συμβόλαια των εργαζομένων που χρησιμοποιούνται ε, για να παρακαμφθεί ο Βρετανικός νόμος που καθορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με παρόμοιο τρόπο, στην περίπτωση του Βέλγιου και των ε, ελαστικών συμβάσεων, οι συμβάσει αυτές εξαιρούν ε, τους μισθούς και μερικές φορές και την ε, ε, αμοιβόμενη ετήσια άδεια από την προστασία που είναι ισχυρή στο Βέλγιο για άλλου τύπου συμβάσεις. Αυτά τα, αυτές οι αδυναμίες στην προστασία των εργαζομένων συνδυάζονται με άλλα κενά στην εκπροσώπηση και στην ε, ε, ε, εφαρμογή. Για παράδειγμα, στα βελγικά, στις βελγικές συμβάσεις οι εργαζόμενοι δεν έχουν δυνατότητα να ε, ισχύσουν για αυτούς ε, αμοιβέ οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο συλλογικών συμβάσεων. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, και στα δύο, στους δύο αυτούς τύπους συμβολέων της, του Ηνωμένου και του Βελγίου ε, δεν χρειάζεται να υφίστανται γραπτός. Αυτό προφανώς δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση των δικαιωμάτων εργαζομένων. Τέλος, τα εθνικά μέτρα σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου δεν αρκούν για να αποφευθούν ε, καταχρήσεις ή να τιμωρήσουν καταχρήσεις που μπορεί να προκύψουν. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι σημαντικό να δούμε πώς το, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά αυτές τις αδυναμίες. Και, ο πρωτογεν, και το πρωτογενές δίκαιο και το δευτερογενές δίκαιο. Το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ερμηνευθεί ως ε, ότι προωθεί υψηλά πρότυπα εργασίας, πρότυπα συνθηκών εργασίας, για όλους τους εργαζόμενους. Αν διαβάσουμε τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των, ε, ανθρωπίνων και το άρθρο 30 για την προστασία από αδικαιολόγητη ε, ε παύση, ε, απόλυση, αυτό εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο τους εργαζόμενους που έχουν ε, στάνταρ συμβόλαια εργασία, αλλά και άτυπα συμβόλαια, μη τυπικά συμβόλαια εργασία. Η πλήρης ισότητα δεν είναι απλώς στόχο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί και γενική αρχή της νομικής τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την νομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να πούμε ότι επανειλημμένω αυτή η νομολογία έχει ε, αποφανθεί για υποθέσεις ε, ισότητας και έχει αποφανθεί ότι ε, η ισότητα στην αγορά εργασίας ε, αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής ε, αξίας και αρχής της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει βέβαια να αξιολογήσουμε και το ε, ε, δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εθνικό δίκαιο. Υπάρχουν, υπάρχουν πρόοδοι. Έχει γίνει πρόοδος μέσω οδηγιών κλπ. Και έχουμε προσπαθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουμε την ισότητα στη μεταχείριση. Για παράδειγμα, οδηγία για την ε, για, για τις συμβάσεις μερικού, μερικής απασχόλησης ή προσωρινού ε, ε, ε, περισμένου χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην, για, στην περίπτωση των συμβάσεων μηδονικού χρόνου. όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν ακόμα Διάφορε αδυναμίε στο δεύτερογενέ δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωση, που ε, έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ε, συνολικής ε, ε, εφαρμογής, της καθολικής εφαρμογής και της ισότητας. Ε, ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ίσως θα μπορούσαμε να το να συζητήσουμε αργότερα το θέμα του δικαστηρίου. Ε, αν μπορεί να μας μιλήσει ο Γιάννης για τα franchise, για τη δικαιόχρηση και μετά θα επανέλθω. Ευχαριστούμε. Και τώρα νομίζω ότι ε, επειδή εσείς ε, χρησιμοποίησα αρκετό χρόνο να δώσω το λόγο σε εσά και θα δούμε τι μελιγενέστε. Μην καθυστερήσουμε και πάρα πολύ. Ένα άλλο τομέα ενδιαφέρον ήταν να δούμε το franchising. Να δούμε δηλαδή ε, τι σχέση υπάρχει μεταξύ του κατακαιρματισμού των επιχειρήσεων και της συλλογική επισφάλειας, βλέποντας τι συνέπειες έχει το franchising, που είναι ένας τρόπος κατακαιρματισμού της εργασίας που χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα του fast food για την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο. Δεν μπορώ να πω πολλά για το πώς ακριβώς ε, δομείται το franchising, αλλά Υπάρχει ένας παράδοξος ε, συνδυασμός νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας όλων. Για παράδειγμα, τα McDonald's, τα Starbucks ε, ως επιχείρηση της οποίας κάποιος αναλαμβάνει το franchise, αλλά υπάρχει και ισχυρή άσκηση ελέγχου από τον ιδιοκτήτη του franchise. Και φυσικά ε, υπάρχει δυνατότητα αυτή του ελέγχου που μπορεί να επηρεάσει και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε επίπεδο franchising. Η πρόκληση είναι κατά πόσον ε, θα πρέπει οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να καθορίζονται σε κάθε μονάδα, δηλαδή σε κάθε κατάστημα McDonald's για παράδειγμα, ή αν θα γίνεται σε επίπεδο δικτύου. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πιστεύουμε ότι το franchising θα πρέπει να θεωρείται ε, ε, ένας ε, παράγων ο οποίος μπορεί να δώσει τη δυνατότητα επισφαλούς εργασίας υψηλού κινδύνου και μπορεί επίσης να αποσυνδέσει την ε, επιχείρηση από τον κατακαιρματισμό. Είναι σημαντικός μηχανισμός επιχειρήσεων, αλλά αυτός ο κατακαιρματισμός της επιχείρησης δεν θα πρέπει να οδηγήσει και σε κατακαιρματισμό ε, στη δυνατότητα να εισακούγεται η φωνή του εργαζομένου. Αυτή η παράπλευρη συνέπεια λοιπόν του ε, franchising σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ε, κεφαλαιοποιούν τη δυνατότητα και είτε αποκλείονται οι εργαζόμενοι τελείως από δομές εκπροσώπησης, ε, εδώ υπάρχουν θέματα ικανοποίησης ή στο κάθε κατάστημα ικανοποιούνται κάποια κατόφλια, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να μην είναι πολύ αποτελεσματικά και δεν μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το εργατικό δυναμικό για την άσκηση των δικαιωμάτων του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της εργασίας μέσω franchising. Αν υπήρχε βέβαια ένα εύρωστο νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς κενά στην εφαρμογή, τότε μπορεί να μην υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, διότι υπάρχει επισφάλεια κυρίως μέσω παραγωγού δικαίου. Το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει ε, ευρύτερα μια στρατηγική κατά τη επισφάλιση, αναγνωρίζει συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα, συλλογικέ συμβάσει, δικαιώμα στην απεργία και δικαιώματα ε, soft law, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα κενά ε, κοινωνικής πολιτικής αρμοδιότητας που αποκλείουν κάποια δικαιώματα. Θα δούμε λοιπόν τέσσερι οδηγίε. Μία οδηγία είναι η οδηγία ε, για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας. Η δεύτερη είναι η οδηγία για τις ε, ε, συλλογικές απολύσεις και ε, τις ε, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Υπάρχουν κάποια κενά, δεν έχω χρόνο να σας πω λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα βεβαιότητας και πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτά ισχύουν και για τα δίκτυα franchising, κατά πόσο μια επιχείρηση ε, στην οδηγία μπορεί να θεωρείται ότι ισχύει και για το δίκτυο του franchising και το ίδιο ισχύει αφορά και τις συλλογικέ απολύσεις. Εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει προβληματικό κενό είναι στην περίπτωση που μεταβιβάζεται η επιχείρηση σε άλλον και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ε, δεν μπορούν ε, να εισακουστούν και να ακουστεί και η δική τους η άποψη κατά τη μεταβίβαση, παρά το γεγονός ότι φύγονται τα δικαιώματά τους. Αυτά φυσικά ε, έχουν να κάνουν και με κενά σε επίπεδο κρατών μελών, πέραν από τα κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δίνουν στη δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, να δούμε τι γίνεται με τους εθνικούς κανόνες ε, εργατικού δικαίου και εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ευρύτερος ορισμός του εργαζομένου ε, που θα ισχύει όπως γίνεται και με θέματα προστασίας. Αυτά τα κενά λοιπόν μπορεί να επιτρέψουν σε χώρες να έχουν περιορισμούς για απεργία ή συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να είναι προς όφελος των δικτύων ε, franchising. Για παράδειγμα, όταν σε μια χώρα απαγορεύεται ε, δευτερογενή απεργία. Δηλαδή, μία απεργία σε ένα κατάστημα McDonald's δεν μπορεί να την υποστηρίξουν εργαζόμενοι σε άλλο κατάστημα McDonald's, που σημαίνει ότι περιορίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το δικαίωμα τη εκπροσώπησή του. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα δίκτυα του franchising για να δούμε κατά πόσον υπάρχει και κατάλληλη ε, εκπροσώπηση. Ε, το άλλο το οποίο εξετάζουμε είναι το θέμα το, ε, των σχέσεων μεταξύ των διαφορών μέτρων πολιτικής. Ε, πρέπει να υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που να είναι σωστές, αλλά αν υπάρχει κάποια η οποία είναι λανθασμένη, μπορεί να υποσκάπτει όλα αυτά τα θέματα της επισφάλειας. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που εντοπίσαμε. Ο πρώτος είναι η αλληλεπίδραση με τον κανονισμό για το χώρο εργασία. Το γεγονό ότι στην οδηγία δεν υπάρχει ένα δικαίωμα για ελάχιστες ώρες εργασία. Όχι μέγιστο, αλλά και ένα ελάχιστο όριο όρων ε, ε, εργασίας ε, μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικέ εργασίες και τελικά στον εργαδότη ο οποίος έχει έλεγχο για το χρόνο εργασία. Ένα άλλο είναι η σχέση μεταξύ άτυπων μορφών εργασία και το δικαίωμα του εργαζομένου να γνωρίζει τις συνθήκες απασχόλησης όπως εκφράζονται στις οδηγίες ε, των γραπτών δηλώσεων. Εδώ υπάρχει μια εθνική διάσταση που αφορά την προσωπική αξιοπρέπεια του ατόμου, να γνωρίζει κάποιο τι δικαιώματα έχει και τι υποχρεώσει. έχει οικονομική λογική, οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ολοκλήρωση αγορά αγοράς και είναι και μια στρατηγική αποτελεσματικότητα γιατί μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία, να παρακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωση με βάση εργατικά πρότυπα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εργάζονται περιστασιακά και δεν καλύπτονται από την προστασία της οδηγίας για τις γραπτές δηλώσεις και θεωρούμε ότι αυτό είναι κενό προστασία, διότι υπάρχει το παράδοξο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που απαιτούν περισσότερο, χρειάζονται μάλλον περισσότερο να μπορούν να στήσουν τα δικαιώματά τους. Και η σχέση μεταξύ του κατακαιρματισμού των επιχειρήσεων στην άτυπη της απασχόλησης και της επισφάλεια έχουν μια σχέση. Ο κατακαιρματισμό μια επιχείρηση, όπω είδαμε, για παράδειγμα σε ένα franchise, σημαίνει ότι μπορούν να δοθούν κίνητρα λόγω της δομής του franchise ε, να υπάρχει μια στρατηγική χαμηλού κόστους για να μειώσουμε το κόστος της εργασίας. Για παράδειγμα σε τομείς όπως είναι τα fast food. Ε, οι εργοδότες μπορεί να έχουν κίνητρο να εφαρμόσουν άτυπες μορφές εργασίας αυτοί οι άτυπα εργαζόμενοι ε, με τη σειρά τους μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορα προσκόμματα όσον αφορά την εκπροσώπησή τους. Αν είσαι ένας εργαζόμενος με, με μια σύμβαση μηδενικών ωρών, επειδή φοβάσαι ότι δεν θα χάσει τη δουλειά σου ή ότι δεν θα έχεις ώρες εργασίας την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να μην βρει τα κίνητρα για να οργανώσεις ε, ε, τα δικαιώμα... και να ασκήσεις τα δικαιώματα εκπροσώπησή σου. Και επειδή δεν υπάρχουν δικαιώματα εκπροσώπης, μπορεί να υπάρχουν ε, δημοκρατικά ελλείμματα στο χώρο εργασία και επομένως δεν μπορεί να αντισταθμίσουν ε, τι αποφάσει του εργοδότη. Όλα αυτά είναι από κοινού και προκειμένου να υπάρχει μια κατάλληλη στρατηγική για αυτά, πρέπει να σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο. Και τώρα θα δώσω και πάλι το λόγο στην Αριστεία για να ολοκληρώσει. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν όσον αφορά τι προτάσει πολιτική. αν το πρόβλημα μεταφοράς του κινδύνου είναι από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, είναι παρεμβατικό και αφορά όλη την αγορά εργασία, θεωρούμε ότι αυτό θέτει βαθιά ερωτήματα για την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να πούμε ότι ο κανονισμός για την αντιμετώπιση τη μεταβίβασης του κινδύνου ε, στο εργατικό δυναμικό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει ολιστικά, διότι υπάρχει ακριβώς αυτή η επισφάλεια που είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται σε διάφορες μεταβλητέ. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε ένα πίνακα με συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής, ε, τις οποίες αναφέρουμε και στην έκθεση και κατ' ουσίαν ε, είναι κατηγοριοποιημένες επί τη βάση τριών αρχών. Καταρχάς, στην αρχή ε, τη έλλειψη αποκλεισμού. Ε, και εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά την εισαγωγή ενός πανευρωπαϊκού ορισμού ε, για τον εργαζόμενο. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για μια σειρά από εργαζομένους που εργάζονται με περιστασιακά άτυπα ε, συμβόλαια για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα εργαζομένων. Μια άλλη πρόταση που είναι ε, πάλι σε αυτό το πλαίσιο της έλλειψης αποκλεισμών είναι να εξορθολογήσουμε το franchising με την οδηγία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση για να υπάρχει εφαρμογή καθολικά σε όλους τους εργαζομένους ε, χωρίς κατακαιρματισμό. Και βεβαίως ε, θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά για λόγους ισότητα, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση πολιτικής όσον αφορά την επισφαλή εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κείμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο στα θέματα της εργασίας, αλλά και στο θέμα τη ρύθμιση του χρόνου εργασία. Όπω συζητήθηκε ε, και στην έκθεση και σήμερα στην παρουσίαση, ούτε η οδηγία για την... Ε, εργασία ε, μερικής απασχόλησης ή η οδηγία για το χρόνο εργασία, ε, δεν καθορίζει κάποιον ελάχιστο χρόνο εργασία που πρέπει να παρέχεται στον εργαζόμενο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθμίσουμε αυτό το κενό, να υπάρχει δηλαδή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες ώρες εργασία οι οποίε θα πρέπει να προσφέρονται στον εργαζόμενο. Και ε, κατόπιν, τέλος, στην ανάλυση μας διαπιστώσαμε ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες πάσχουν και από κενά στην εφαρμογή τους. Και θεωρούμε ότι, όπως είπαμε και στην έκθεση, υπάρχουν μια σειρά από συστάσεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Καταρχάς, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες ε, που αφορούν την απασχόληση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ε, τροποποίησης της οδηγίας για τις γραπτές δηλώσεις ε, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τη μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για την προστασία των εργαζομένων. Εδώ υπάρχουν διδάγματα, για παράδειγμα, ε, ε, τα οποία θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε από την νομοθεσία περί διότι καλύπτουν και κάποια προστασία όσον αφορά τη θυματοποίηση κλπ. Ε, ολοκληρώνοντας βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί, θεωρούμε, εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι ίδιοι και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες δεν κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουν τα θέματα της επισφάλειας και να φροντίσουν να προωθήσουν εργασία η οποία θα συνάδει με τους στόχους της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και ε, της έλλειψης αποκλεισμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Η μελέτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε που περιγράψατε τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Τώρα θα δώσω το λόγο σε συναδέρφους για να θέσουν ερωτήσεις προς τους δυο σας. Jude. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έχασα το ξεκίνημα της παρουσίασης και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν ήδη έχει καλυφθεί η ερώτησή μου. Στα συμπεράσματά σας αναφερθήκατε στο ότι ένα από τα συμπεράσματα της μελέτης ε, είναι τα κενά ε, στην νομοθεσία. Για να καλυφθούν αυτά, μπορεί κανείς να νομοθετήσει ή να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία. Προφανές είναι ότι δεν έχει υπάρξει κοινωνική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, εδώ και πάνω από μία δεκαετία και πολλά και υπάρχουν κενά και ε, το εργασιακό δίκαιο δεν έχει εξελιχθεί με, στον ίδιο ρυθμό με τις εξελίξεις ε, στην αγορά εργασίας. Ε, λοιπόν, μπορεί κανείς αφενός να νομοθετήσει για να καλύψει τα κενά ή να καλυφθούν τα κενά μέσω της νομολογίας, μέσω των δικαστηρίων. Στα συμπεράσματά σας αναφέρεστε στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και μου φαίνεται ότι μία από τις ε, μεγαλύτερες δυσκολίες ε, για ε, τους εργαζομένους σε άτυπες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης όποιο και αν είναι το σύστημα του κράτους μέλους, το θέμα είναι εάν είναι ανοιχτό το σύστημα αυτό για την πλειοψηφία των ανθρώπων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ισχύει αυτό λόγω του ύψους των τελών. Αλλά ακόμα και αν είναι υπάρχει κίνδυνος για τον εργαζόμενο εάν προσφύγει. Και αυτό είναι τεράστιο βάρος ε, για ένα άτομο ή για μια μονάδα ατόμων. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, κατά τη γνώμη σας, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν νομοθετήσουμε, που θα ήταν η πρώτη μου προτίμηση, να βελτιώσουμε δηλαδή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να καλύψουμε τα κενά, τα παραθυράκια που υπάρχουν και να φροντίσουμε το δίκαιο για την απασχόληση να ακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία. Ε, εάν δεν το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να φροντίσουμε οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους ε, να ε, μπορέσουν να σπρώξουν, να ασκήσουν πίεση για να κλείσουν τα κενά. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πρόεδρος, ε, αναφερθήκατε και στο κενό όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Ε, ε, αυτό λοιπόν προστίθεται στην ερώτηση της Τζούντ. Παρακαλώ. Ναι, καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε και είναι αλήθεια ότι τέτοιου είδους κενά που έχουμε, εντυπώσει, που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στην αλλαγή πρακτικών Συμφωνούμε λοιπόν με τη δική σας ερμηνεία όσον αφορά το πού προέρχονται τα κενά αυτά. Όσον αφορά τη δυνατότητα νομοθεσίας και έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αυτή θα μπορούσε να είναι μια πιθανή οδόση για τροποποίηση της νομοθεσίας. Ε, υπάρχουν προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο για πολιτικούς αλλά και νομικούς λόγους να νομοθετήσει κανείς και να τροποποιήσει την νομοθεσία σε όλους τους τομείς που έχουμε εντοπίσει. Εάν ε, ισχύει αυτό, τότε ε, άλλος δρόμος που θα μπορούσε να ακολουθηθεί είναι να υπάρχουν ε, καλύτεροι μηχανισμοί επιβολής του νόμου και να παρακολουθείται η εφαρμογή από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κρατών μελών. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ε, κάποια κενά που, που διαπιστώσαμε συγγνώμη, οφείλονται σε ελλειπή εφαρμογή κάποιων οδηγιών. Διαφορετική διαδικασία λοιπόν θα μπορούσε ενδεχομένω να παράσχει έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση αυτών των κενών. Άλλο θέμα που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η εκπροσώπηση, να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων, να υπάρξει μηχανισμός για να καλύψουν για να καλυφθούν τα κενά. Αλλά το πρόβλημα και πάλι για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι και αυτό είναι κάτι που δεν ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω εάν ο Γιάννης έχει κάτι να προσθέσει σε αυτά. Πολύ σύντομα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι, να διαπιστώσουμε ότι η επισφάλεια είναι σημαντική πρόκληση και χρειάζεται καινοτόμε και δημιουργικές λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι οι κοινωνικοί εταίροι να συζητήσουμε. Να συζητήσουν. Έχουμε υποβάλει την πρόταση, υπάρχει και η οδηγία πλαίσιο για τις ε, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Φυσικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή απαιτώνται καινοτόμες λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, δεν είναι? Λίγες μέρες ε, μόλις μετά τη συζήτηση του κοινωνικού πυλώνα στο Γκέτεμπορκ, στη Σουηδία, ε, συζητάμε το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει κανονισμός, ε, δεν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση και τα κράτη-μέλη δεν θέλουν πλήρη εναρμόνιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Δεν είμαστε ομοσπονδία, είμαστε συνομοσπονδία κρατών. Και τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητες ε, στον τομέα αυτών. Ε, θα πρέπει λοιπόν με πολύ προσοχή ε, να κινηθούμε και να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησης, το πρώτο πάνελ, ε, θα ασχοληθεί με τις επισφαλές συνθήκε εργασία στην Ευρώπη το 2017. Ε, με χαρά καλωσορίζω τον ε, συντονιστή της συζήτησης, τον συνάδελφο και πολύ αγαπητό φίλο, Χάιν Μπέκερ, που θα προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ. Θα με συγχωρήσετε που πρέπει να αποχωρήσω. Θα επανέλθω το συντομότερο δυνατό. Κύριε Μπέκερ, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καλωσορίσατε στο πρώτο πάνελ, στο πρώτο τμήμα της ε, σημερινής ακρόασης. Ε, είμαι προβλεφτής από το 2011 και έχω την τύχη να ε, συμμετέχω στην Επιτροπή Αναφορών ως μέλος και είμαι αναπληρωτής στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πολύ χαίρομαι λοιπόν ε, που ε, ε, έχω εικόνα και των δύο πλευρών αυτών. Στο πρώτο πάνελ θα ακούσουμε τις απόψεις εκπροσώπων ε, Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομάδας Προβληματισμού και Επιμελητηρίου. Και τέλος, θα ακούσουμε τις απόψεις του εισηγητή της έκθεσης για τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση. Στόχος είναι να εξετάσουμε την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, πολύ σωστά μόλις είπε η Πρόεδρος. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που έχει να κάνει με τις ε, εξελίξεις όσον αφορά την διαφοροποίηση των ε, συνθήκων εργασίας. Υπάρχουν οι συμβάσεις μηδενικού χρόνου, υπάρχουν οι ευέλικτες συμβάσεις, ε, οι συμβάσεις flexi time. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και μια άλλη εξέλιξη. Όπως όλοι γνωρίζουν, ε, αυτή είναι η ε, ψηφιοποίηση της οικονομίας που αναδιαμορφώνει τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων βρισκόμαστε εν μέσω της πρώτης φάσης ψηφιοποίησης και όπως όλοι γνωρίζουν, οι συνθήκες εργασίας δεν έχουν ακολουθήσει απολύτως τις εξελίξεις. Ήδη σε πολλούς ε, τομείς της οικονομίας βλέπουμε τεχνολογικές αλλαγές που φυσικά προσφέρουν πολλές ευκαιρίες, ε, φέρουν όμως και πολλές προκλήσεις μαζί τους. Ε, από την χθεσινή συζήτηση συγκράτησα τον όρο «Η νέα ψηφιακή εποχή 5.0». διότι η ψηφιοποίηση αλλάζει τον τρόπο ζωής και εργασίας μας ε, και η ψηφιακή επανάσταση, όπως είπα, φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση της ισορροπίας ε, ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας ε, για όλους, ε, κάνει την αγορά εργασίας ε, πιο ανοιχτή σε όλους. Χρειάζονται όμως μεταρρυθμίσεις. οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα στα κράτη-μέλη. Και γιατί αναφέρομαι στα κράτη-μέλη, διότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταρρυθμίσεων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. το σύνολο της επαγγελματικής κατάρτισης δεν ε, είναι προσαρμοσμένο στη νέα εποχή. Θα υπάρξουν νέα επαγγέλματα, δεν ε, καλύπτονται όμως από την επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχουν κάποιες ε, καλές πρακτικές, δεν τις βλέπουμε όμως παντού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς και όπως αναφέρεται και στην ε, μελέτη, συχνά η εφαρμογή των ε, μέτρων ε, δεν γίνεται εγκαίρος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι πάντα ζήτημα νέας νομοθεσίας, αλλά ζήτημα έγκαιρης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Και θα πρέπει να εξετάσουμε ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, την ενημέρωση των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών και δεν αποτελεί αυτό αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν μια πολύπλοκη κατάσταση όπως ήδη αναφέρθηκε και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες εξελίξεις. Εάν δεν είναι το καταλληλότερο μέσο η νομοθεσία, τότε θα πρέπει να ασκήσουμε ήπια πίεση από πλευρά ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να έχουμε μη δεσμευτικά μέτρα. Αυτές λοιπόν είναι οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις και περνούμε τώρα στους ομιλητές που ελπίζουμε να παρουσιάσουν τις να μας παρουσιάσουν τα στοιχεία τους εντός 10 λεπτών. Ελπίζω να μπορέσουν να ε, περιοριστούν. Ε, εάν όχι, θα ακούσετε εδώ το καμπανάκι. Κατόπιν ε, θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Καλωσορίζω λοιπόν τώρα τους εξής ομιλητές, την Ιζαμπέλα Μπιλέτα, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση ε, των ε, Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας από την Ιρλανδία. Κατόπιν έχουμε την κυρία Ίγκα Μάγτα, Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου ε, Διαρθρωτικών Ερευνών από την Πολωνία. Έχουμε τον Ρολφ Γκλάισνερ, αναπληρωτή διευθυντή κοινωνικής πολιτικής ε, στο Αυστριακό Επιμελητήριο. Εκπροσωπεί δηλαδή από την πατρίδα μου την Αυστρία, τους κοινωνικούς εταίρους από την πλευρά των ε, εργοδοτών. Και τέλος έχουμε τον Νεοκλή Σιλικιώτη, συνάδελφο εδώ από το Ευρωκοινοβούλιο, εισηγητή της έκθεσης ε, για τη συνθήκη εργασίας και την επισφαλή απασχόληση από την Επιτροπή Απασχόλησης. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπιλέτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλη την Επιτροπή Αναφορών που ζήτησε από το Eurofound να συνεισφέρει σε αυτή τη δημόσια κρόση ένα θέμα το οποίο το έχουμε εξετάσει από πολλές οπτικές γωνίες. Για, σε σχέση με τις επισφαλείς συνδέξεις εργασίας, με τα, τις άτυπες μορφές εργασίας, τις απα, ε, απατηλές μορφές εργασίας, ε, τις παράνομες δηλαδή μορφές εργασίας κλπ. Ας δούμε λοιπόν τι είναι η επισφαλής εργασία και η επισφαλής απασχόληση, η επισφαλής συνθήκες εργασίας. Όπως είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, εδώ ε, επικρατεί μια πραγματική αβεβαιότητα ακόμα και σε ό,τι αφορά τον ορισμό. Κατά κάποιο τρόπο η επισφαλής απασχόληση περιγράφεται συνήθως αρνητικά. Δηλαδή μια σχέση εργασία που δεν είναι παραδοσιακή. Δεν είναι δηλαδή μόνιμη, πλήρης ε, απασχόληση ανάμεσα σε ένα εργαζόμενο και ένα εργοδότη. Όπως και άλλοι ε, ερευνητές, ε, ο Ριμ και ο Ρούμπερι έχουν πει, μιλούμε για σχέσεις εργασίας οι οποίες δεν προστατεύουν τον εργαζόμενο, δεν επιτρέπουν στον εργαζόμενο να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα ε, τα οποία θα του έδινε μια καλή θέση εργασίας. Μιλώντας για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ταυτόχρονα και την ποιότητα εργασίας, την ποιότητα της απασχόλησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διευρύνουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σήμερα. Γιατί, γιατί οι θέση θέσεις απασχόλησης δεν είναι απλώς μια άτυπη μορφή εργασίας. Συνδέεται και υφίσταται ακόμα και στις συνήθεις ε, παραδοσιακές σχέσεις εργασίας. Και θα επανέλθω σε αυτό. Αυτό είναι το περιεχόμενο το οποίο θα διατρέξω εντάχει. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τα χαρακτηριστικά της επισφαλούς εργασίας και κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους αυξάνεται η επισφάλεια και για μερικούς από τους λόγους για τους οποίους αυξάνεται η επισφάλεια καθώς επίσης θα μιλήσω και για τις βασικές προκλήσεις. Καταρχήν για τα χαρακτηριστικά. Να σας δείξω αυτό εδώ το είναι εδώ τη διαφάνεια για να σας δείξω τι έχουμε κάνει εμείς στην επισκόπηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών Εργασίας που έκανε το Eurofound. Ε, κάνει το Eurofound εδώ και 25 χρόνια, κάθε πενταετία. Ε, σε όλη την Ευρώπη ρωτάμε τους εργαζόμενους ποια είναι η εμπειρία τους από την εργασία τους, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας τους. και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν εξετάσουμε μια σειρά από παράγοντες και από διαστάσεις που συνδέονται και με την επισφάλεια. Η επισφάλεια δεν αφορά μόνο ένα χαρακτηριστικό, είναι μια σειρά παραγόντων οι οποίοι τη δημιουργούν. Οπότε ακόμα και στις συνήθεις παρουσιακές σχέσεις εργασίας μπορεί να υφίσταται επισφάλεια όταν εξετάσουμε όλους τους παράγοντες. Ε, εξετάζουμε τα ε, προφίλ της ε, ποιότητας εργασίας με βάση πέντε χαρακτηριστικά. το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος, ε, ένταση εργασίας, ποιότητα του χρονοεσίας, ε, προσδοκίες ε, και ε, μισθή. καθώς επίσης και τα, τις ικανότητες που χρειάζονται και που χρησιμοποιούνται. Αυτό που βλέπετε σε αυτό το γράφημα είναι ότι έχουμε ένα, μια ποικιλία ποιότητας εργασίας και δεν μιλούμε μόνο για τις άτυπες μορφές εργασίας. Έχουμε ε, μια πολυμορφία στην ποιότητα. Βλέπουμε ε, 13%, 19% και 22% των ε, από το 13% εν πάση περιπτώσει μέχρι το 25% ε, ανάλογα με το δίκτυ είναι θέσεις εργασία χαμηλής ποιότητας. Το 1 τρίτο των εργαζομένων βρίσκονται σε προφίλ θέσεων εργασία χαμηλής ποιότητας και εκφράζουν φόβους να απολέσουν τη θέση τους στους επόμενους 6 μήνες. Υπάρχει πολύ χαμηλή χρήση προσόντων και πολλούς και πολύ υπερβολικά πολύ νέοι με λίγα προσόντα σε αυτές τις χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Να δούμε, ε, για παράδειγμα, την ένταση εργασίας. Ακόμα και για να αξιολογήσουμε αυτό μόνο τον παράγοντα, χρειάζεται να τον κατατμήσουμε σε διάφορα στοιχεία. Για παράδειγμα, εργασία σε υψηλή ταχύτητα, ε, η ε, παράγοντες ε, που δυσχεραίνουν την εργασία κλπ. Υπάρχουν ε, παράγοντες οι οποίοι ε, επηρεάζουν αυτές τις διαστάσεις και επηρεάζουν και την ποιότητα εργασίας λοιπόν. Δεύτερο σημείο το οποίο μου ζητήθηκε να εξετάσω είναι οι ε, παράγοντες οι οποίοι επιτείνουν την επισφάλεια. Ε, αυτό το γράφημα δεν είναι πολύ σαφές όταν το βλέπει κανείς, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας σε ό,τι αφορά το καθεστώς της ε, απασχόλησης αυτή τη στιγμή. επειδή αυτή την επισκόπηση, αυτή την επισκόπηση την κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τι έχουμε, πού έχουμε καταλήξει. Πηγαίνουμε και ρωτάμε τους εργαζόμενους στο χώρο εργασία τους ε, ποιο είναι το καθεστώς με το οποίο εργάζεστε. Βέβαια τους το λέμε έτσι. Τους λέμε είσαστε ε, εργαζόμενος, απασχολούμενος κλπ. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν μπορούν να πούν ότι είναι αυτοπασχολούμενοι ή μισθωτοί. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε επιμέρους ερωτήσεις για να διαπιστώσουμε πού θα πρέπει να ταξινομηθεί ο κάθε εργαζόμενος. Βλέπετε εδώ, του ρωτάμε, πληρώνεστε μισθούς, πληρώνεστε επιδόματα, ε, ε, είσαι αυτοπασχολούμενος, εργάζεσαι για τον εαυτό σου ανεξάρτητος εργαζόμενος. Ε, ακόμα και, και πάλι όμως <laughs> δεν έχουμε τη δυνατότητα να ταξινομήσουμε όλους τους εργαζόμενους. Δεν μπορούν οι ίδιοι να ταξινομήσουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακόμα υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή την ε, μη σαφή διάκριση ανάμεσα στους αυτοαπασχολούμενους που ε, εμπίπτουν στο εμπορικό ή στο αστικό δίκαιο και τους μισθωτούς που εμπίπτουν στο εργατικό δίκαιο. Μετά, να δείτε εδώ πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ακριβώς την αυτοπασχόληση. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι ακριβώς τα κριτήρια τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι οι αυτοπασχολούμενοι είναι πραγματικοί αυτοπασχολούμενοι και όχι ε, ε, ε, πραγματικά στην πράξη μισθωτή. Για παράδειγμα, αν έχουν μόνο ένα ή περισσότερους εργοδότες, αν έχουν ε, τη δυνατότητα να λαμβάνουν οι ίδιες στρατηγικές αποφάσεις ε, για την εργασία τους κλπ. Τότε είναι αυτοαπασχολούμενοι. Αν όμως αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται ή πληρείται μόνο ένα, τότε ο εργαζόμενος είναι μάλλον εξαρτώμενος, ενδεχομένως μισθωτός αν δύο από τα κριτήρια πληρούνται και όχι τα υπόλοιπα, βρίσκεται κανεί σε μια γκρίζα ζώνη, στην οποία πραγματικά δεν ξέρουμε πού να κατατάξουμε τον εργαζόμενο και εκεί είναι σημαντικό ότι θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί μέσω νομοθεσίας. Το θέμα της ε, αυτοαπασχόλησης, ε, της ψευδούς αυτοπασχόλησης ή της ε, μισθωτής εργασίας έχει αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα τρίτο καθεστώς ad hoc που είναι ανάμεσα στο, στη μισθωτή εργασία και την αυτοπασχόληση. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αργότερα γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Το τρίτο σημείο, τρίτος παράγοντας που επιτείνει την επισφάλεια είναι αυτό που είπατε και εσείς Πρόεδρε για τις ε, νέες μορφές εργασίας οι οποίες προκύπτουν. Θέλω να επιστρέψουμε στο καθεστώς και των εργοδοτών, όχι μόνο των αζωμένων. Τι είχατε πει εσείς? για, τις, ε, για τη δικαιώξη πέραν της, ε, των franchise. Ε, γιατί έχετε, επειδή έχετε τους αποσπασμένους εργαζόμενους, ε, δημιουργείται η απόλυτη διάκριση ανάμεσα ε, τις ε, διάφορες λειτουργίες του εργοδότη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει, ποιος είναι αυτός ο οποίος προσλαμβάνει, ποιος είναι αυτός που απολύει. Μπορεί να είναι διαφορετικοί αυτοί οι άνθρωποι, οι οντότητες. Οπότε έχουμε επισφάλεια και επισφαλείς συνθήκες εργασίας όχι μόνο στις άτυπες μορφές εργασίας, αλλά και στις στάνταρ στις παραδοσιακές, τυπικές μορφές εργασίας. Για παράδειγμα, 22% των εργαζομένων εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους προκειμένου ε, να καλύψουν τη ζήτηση ή 26% εργαζομένων που δεν, δεν ε, ξεκουράζονται για 11 ώρες τουλάχιστον μεταξύ δύο ε, εργάσιμων ημερών. Τέλος, οι βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Πρώτον, η συνεχώς αυξανόμενη μεταφορά κινδύνων στους ε, εργαζόμενους. Επίσης δεν μιλήσατε εσείς για τα κενά στο συστήματα κοινωνικής προστασίας. Υπάρχουν κενά στα συστήματα ε, κοινωνικής προστασίας και αυτό είναι ένας ε, παράγοντας που επιτείνει την ε, επισφάλεια. Τα συνδικάτα πρέπει να μπορούν επίσης να εκπροσωπούν όχι μόνο τις εργαζόμενους σε άτυπες μορφές εργασίας, αλλά και τους επισφαλείς εργαζόμενους. Και αυτό είναι μια πρόκληση για το, τα συνδικάτα, πρόκληση νομιμοποίησης. Ε, Επίσης, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ε, είναι και αμοιβόμενοι εργαζόμενοι και μη αμοιβόμενοι εργαζόμενοι ταυτόχρονα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε την προοπτική στο μέλλον. Για παράδειγμα, οι γυναίκες δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιληφθούν το μέλλον τους. Δηλαδή, αν χάσουν το, ε, το καθεστώς ε, του εργαζόμενου όταν αποκτήσουν παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσουν ξανά στο μέλλον. Επίσης, ε, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ε, ε, πίπεδο της, της Ευρωπαϊκής γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κατευθύνσεις οι οποίες θα ε, δώσουν, στις οποίες θα οικοδομήσουν τα κράτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Eurofound ε, πλήρει τις προσδοκίες. Να καλωσορίσουμε αρκετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους συναδέλφους μου εδώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον ε, στο θέμα, για το θέμα αυτό. Η κυρία Μάγκτα τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. 10 ή 15 λεπτά έχω στη διάθεσή μου. 15, ωραία. Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο στόχος μου είναι να σας δώσω μία σύντομη εισαγωγή για την κατάσταση στην αγορά εργασίας της Πολωνίας με στόχο να σας παρουσιάσω πώς ε, η δική μας η δομή της αγοράς εργασίας άλλαξε τις τελευταίες δύο δεκαετίες ε, όσον αφορά τις διάφορες μορφές απασχόλησης. Πρόκειται για μία διαφάνεια εδώ που σας δείχνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας και τη δομή ε, των θέσεων εργασίας που άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Το 2002 είχαμε μια πολύ καλή κατάσταση με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, πάνω από 20% τότε. Αυτό βελτιώθηκε ουσιαστικά έκτοτε με το ποσοστό της ανεργίας να πέφτει στο 5% πλέον αλλά στο μεταξύ μεγάλος αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν τότε ήταν ε, προσωρινής απασχόλησης ε, βλέπετε εδώ το ανοιχτό ροζ, αυτό είναι εκατομμύρια θέσεις εργασίας που είναι προσωρινές ε, θέσεις απασχόλησης. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο περίπου το 2002 και τώρα έχουμε αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια. Ε, διπλασιάστηκε και παραπάνω δηλαδή μέχρι το 2015. Πάνω από το 86% λοιπόν της καθαρής αύξησης της απασχόλησης εκείνο το διάστημα διαπιστώθηκε σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. τίνουμε λοιπόν να λέμε ότι η Πολωνία έγινε μια δεύτερη Ισπανία. Η Πολωνία σε κάποια χρόνια ξεπέρασε την Ισπανία όσον αφορά το μερίδιο της προσωρινής απασχόλησης. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που δείχνει τη ε, ε, σχέση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλο μερίδιο προσωρινής απασχόλησης σε κάποιες χώρες, ιδίως για την Πολωνία εδώ τμήμα της δημιουργίας των θέσεων εργασίας οφείλεται ή παρατηρείται λόγω της αύξησης της ε, παρουσίας ε, υπηρεσιών, ε, ε, οργανισμών που παρέχουν θέσεις προσωρινής απασχόλησης, εταιριών συγγνώμη, που παρέχουν θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Αυξήθηκαν λοιπόν αυτές κατά πολύ στο διάμεσο διάστημα. Οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης τείνουν να είναι και άνισα κατανομημένες όσον αφορά τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Εδώ λοιπόν στο διάγραμμα βλέπετε το μερίδιο ε, προσωρινών και μόνιμων ε, θέσεων απασχόλησης. Η ε, ροζ είναι οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης, το σκούρο κόκκινο είναι οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης, είτε γιατί το επιθυμούν και κάποιοι εργάζονται ε, με θέσεις απασχόληση που ισχυρίζονται ότι δεν είναι δική του επιλογή, τείνουν να υποεκπροσωπούνται και κατά πάσα πιθανότητα εργάζονται και σε θέσεις απασχόλησης ε, χαμηλών μισθών. Υπάρχουν ε, όλο και λιγότερες υψηλόμισθε θέσει. οι περισσότερες είναι μόνιμε θέσεις απασχόλησης με υψηλού μισθού. Κάποιες νομικές πληροφορίες, έχουμε δύο κατηγορίες προσωρινής απασχόλησης ε, στην ε, Πολωνία. Έχουμε τα, ε, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ε, ρυθμίζονται από το εργατικό δίκαιο και η διαφορά με, από τις σχέσεις συμβάσεις αορίστου χρόνου, που είναι οι μόνιμες συμβάσεις αν θέλετε, είναι καταρχάς η περίοδος κοινοποίησης απόλυσης, που είναι πολύ μικρότερη, είναι δύο εβδομάδες συνήθως, σε αυτή την περίπτωση και επίσης η λήξη του σύμβασης μπορεί να γίνει χωρίς καμία αιτιολόγηση. Ενώ ε, θεωρητικά τουλάχιστον χρειάζεται κάποιος, ε, κάποια αιτιολόγηση για μια σύμβαση ορίστου χρόνου. Ε, και φυσικά επίσης αυξήθηκε και ο αριθμός των λεγόμενων συμβάσεων ιδιωτικό δικαίου είναι θέσει των προσωρινής απασχόλησης που δεν προβλέπονται από το εργατικό δίκαιο, ρυθμίζονται από το αστικό κώδικο και δεν είναι τα συνήθη συμβόλαια ορισμένου χρόνου. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπου λοιπόν που έχουμε πλέον συμβάσεις αστικού δικαίου που είναι ε, το μεγάλο ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης. Γιατί είναι τώρα τόσο δημοφιλείς αυτές οι συμβάσεις. Καταρχάς είναι πολύ εύκολο να διακοπούν ανα πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται καμία κοινοποίηση, δεν ε, πληρώνεται αποζημίωση, όλα αυτά φυσικά μετρούν γιατί είναι επιπλέον ε, έξοδα και ε, σχετίζονται και με πολύ μικρότερο φορολογικό κόστος ε, ή δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική εισφορά ή μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλή, ε, ιδιαίτερα σε σύγκριση με συνήθεις ε, συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης και μάλιστα μέχρι το 2016 δεν υπήρχε δέσμευση για κατώτατο μισθό. Η νομοθεσία κατώτατο μισθού που υπάρχει από το 2003 και μετά στην Πολωνία δεν αφορά αυτές τις συμβάσεις σε καμία περίπτωση. Από το 2016 και μετά αφορούν τμήμα αυτών των συμβάσεων αστικού δικαίου. Ε, εδώ έχω ένα πίνακα ο οποίος προσπαθεί να συνοψίσει αυτές τις μορφές ε, συμβάσεων στις πρώτες δύο στήλες έχετε ε, τη συμβάση εργατικού δικαίου που μπορεί να είναι ε, συμβάσει ορίστου χρόνου και συμβάσει ορισμένου χρόνου ε, και όπως σας είπα είναι λίγο πολύ ίδιες. Οι διαφορές είναι κυρίως όσον αφορά την περίοδο κοινοποίησης απόλυσης και την αιτιολόγηση για τους λόγους της απόλυσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ε, ε, ασφαλιστικές εισφορές, κατόπατος μισθός, ισχύει η ίδια νομοθεσία και για τις συμβάσεις ορισμένου και ορίστου χρόνου. Είναι λοιπόν ε, συγκεκριμένες συμβάσεις εργατικού δικαίου και αυτές διαφέρουν από τις άλλες μορφές που σας ανέφερα. Υπάρχει δηλαδή ένας επιπλέον κατακαιρματισμών, υπάρχει η λεγόμενη σύμβαση εντολής, έτσι την μεταφράζουμε από τα πολωνικά, ε, ή συμβάσεις για κάποια συγκεκριμένη εργασία. Ε, προμήθεια, για παράδειγμα, για να γράψει κάποιο ένα βιβλίο. Θεωρητικά αυτές θα πρέπει να είναι οι συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις συμβάσεις αστικού δικαίου, αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για σύμβαση για επισκευές ή για καθαρισμό ε, ακόμα και αν φαίνεται τελείως παράλογο όλο αυτό. Ε, εδώ η διαφορά είναι ότι υπάρχει τελείως ε, διαφορετική ε, αντιμετώπιση σε σχέση με τη συμβάση του εργατικού δικαίου. Καταρχάς, ε, εδώ και κάποιο διάστημα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά ασφαλιστικές εισφορές, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλές, αλλά υπάρχουν και κάποια παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν να αποφύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ε, δεν υπάρχει καμία κάλυψη λοιπόν ε, ασφαλιστικών εισφορών ε, στις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά την αμοιβόμενη άδεια μπορεί να υπάρχει στη σύμβαση κατόπιν συμφωνία. Συνήθως βέβαια έχουμε ελάχιστε συμβάσεις με τέτοιες συμφωνίες που καλύπτουν και πληρωμένη άδεια. από το 2016 υπάρχουν κάποια διαμεστικά στοιχεία για τις ε, ε, συμβάσεις εντολής όπως τις αποκαλούμε. Υπάρχει ένα ελάχιστο όριο εργασιών ημερήσιο, αλλά υπάρχουν και νέοι τρόποι να παρακάμψουμε όλα αυτά ε, στον κανονισμό. Και φυσικά ε, δεν υπάρχει καμία περίοδος κοινοποίησης ε, στις συμβάσεις αυτές. Ε, βεβαίως μπορεί στο σύμβαση να συμπεριληφθούν κατόπιν συμφωνίας. Δεν χρειάζεται να δοθεί καμία αιτιολόγηση για την διακοπή της σύμβασης, δεν ε, καταβάλλεται αποζημίωση για να κάνει κάποιος κάτι συγκεκριμένο και ε, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ε, στις συμβάσεις αυτές της εντολής, contracts of mandate όπως αποκαλούνται. Καταρχάς αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κενά για την κοινωνική ασφάλιση των ε, εργαζομένων και την κοινωνική τους προστασία, ε, πρόσβαση κυρίως ε, σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές εισφορές και φυσικά και πολύ σημαντική όσοι είναι ο αντίκτυπος για τα μελλοντικά κενά που θα υπάρχουν στις συντάξεις. Ε, και φαίνεται να υπάρχει και σημαντικός ε, μοχλός αύξησης, ιδιαίτερα σε αυτές τις ε, συμβάσεις αστικού δικαίου. Έγιναν και κάποιες μελέτες που εξετάζουν την ποιότητα και τη διαφορά στην ποιότητα εργασίας. Να παραπέμψω και στη μελέτη της Eurofound και να αντλήσαμε και κάποια διδάγματα από εκεί για το τι γίνεται με αυτές τις συμβάσεις στην Πολωνία και εδώ έχουμε μια πολύ σύντομη επισκόπηση του τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις μορφές συμβάσεων. Ε, όπως είναι λογικό, αυτοί που εργάζονται με αυτά τα ε, προσωρινές συμβάσεις συνήθως έχουν χαμηλότερη ποιότητα εργασίας και αυτό αφορά όλες τις διαστάσεις της ποιότητας εργασίας που εξετάσαμε, ε, δηλαδή χαμηλότερη μισθού, ε, χαμηλότερα κέρδη γενικότερα, υψηλότερο κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους, ε, κακή ποιότητα προγραμματισμού στην εργασία, μεγαλύτερο άγχος, πολύ περισσότερες περιπτώσεις οι οποίες εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ε, δεν υπάρχει πολλές φορές διάκριση από τους εργαζόμενους με σύμβαση αρίστου χρόνου και υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Ε, συνήθως ε, γιατί κάποιοι που είναι νέοι και μόλις εντάσσονται στην αγορά εργασίας ε, εργάζονται συνήθως ε, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και επομένω έτσι ενθαρρύνεται και συμμετοχή σε επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση, αλλά αν το συγκρίνουμε με άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό της επιμόρφωσης και είναι τεράστια η διαφορά. Αυτό για να σας δείξω και ένα διάγραμμα. Εδώ έχουμε μία από τις διαστάσεις της διαφοράς που υπάρχει στην ποιότητα των θέσεων μεταξύ ορίστων ε, συμβάσεων αορίστου χρόνου και ε, προσωρινών θέσεων απασχόλησης. Εδώ έχουμε τις διαφορές ε, το 2005 και το 2010 και 2015. Βλέπετε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό, αλλά αυξήθηκε πολύ μεταξύ του 2010 και του 2015. Για να συνοψίσω λοιπόν, εν συντομία, στην Πολωνία έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωπους οι οποίοι εργάζονται με θέσεις προσωρινής απασχόλησης και Έχουμε 13 ε, περίπου εκατομμύρια εργαζομένους, ε, υπάρχουν μεγάλο ποσοστά επισπάλειας λοιπόν για αυτούς τους 3 εκατομμύρια εργαζομένους και γενικότερα χαμηλότερη ποιότητα στη θέση εργασίας τους. Ε, Όσον αφορά όμως ε, τις ε, θέσεις αορίστου χρόνου και τις θέσεις ε, ορισμένου χρόνου που καλύπτονται από το εργατικό δίκαιο, εκεί δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις κοινωνικές εισφορές, στις ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Η μεγάλη διαφορά είναι με τις θέσεις απασχόλησης που έχουμε εντός των θέσεων προσωρινής απασχόλησης και καλύπτονται από τον αστικό κώδικα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μάγδα θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα ενημερωτική παρουσίαση και αν δεν σας πειράζει θα ήθελα να την παραδώσω αυτή την παρουσίαση μαζί με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις ε, στα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης, διότι είναι αρκετά ενημερωτικός ο τρόπος με τον οποίο μας την παρουσιάσατε. Ε, ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γκάισνερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you. My σας ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά. Ε, είναι οι διαφάνειες. Εγώ θα σας κάνω την παρουσίαση όμως στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω εδώ και την ε, οπτική των επιχειρήσεων. Θα σας παρουσιάσω κυρίως ε, τις εμπειρίες της Αυστρίας, αλλά θα εξετάσω και ε, τα πράγματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αμφισβητήσω κάποιους μύθους με στοιχεία. Θα ξεκινήσω λοιπόν ε, με το ερώτημα αν οι άτυπες ε, μορφές εργασίας ε, είναι ε, ακούσεις ή όχι. Εδώ βλέπετε μια διαφάνεια που αφορά την Αυστρία. Πάνω-πάνω βλέπετε τους άεργους που έχει μειωθεί, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί από το 29% στο 24% τα τελευταία χρόνια και από κάτω βλέπετε τους άνεργους τους ε, αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ε, μονίμους, ε, τους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης και πλήρους απασχόλησης. Βλέπετε λοιπόν ότι το 39 έως 40% των εργαζομένων εργάζεται με πλήρη απασχόληση. Ε, η μόνη μορφή άτυπης απασχόλησης που έχει παρουσιάσει αύξηση στην Αυστρία είναι η μερική απασχόληση. Ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτήν την ε, διαφάνεια την έχω από μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου βλέπετε τα ποσοστά για τις διάφορες μορφές εργασίας. Ε, το 59% των εργαζομένων είναι απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί. Και αν εξετάσουμε τα, τις άλλες μορφές ε, απασχόλησης, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση ή ε, διατήρηση του ποσοστού. Μόνο στην μερική απασχόληση βλέπουμε αύξηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά είναι από την μελέτη της Eurofund που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μόνη κατηγορία άτυπη μορφής απασχόλησης που έχει ε, αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ύφεση ε, είναι η μερική απασχόληση. Το άλλο που ακούει κανεί ε, συχνά είναι ότι οι άτυπε μορφέ εργασίας είναι επισφαλεί επισφαλής απασχόληση και ότι συνδέονται με την φτώχεια ή με τον κίνδυνο για φτώχεια. Αυτό ισχύει. Στην Αυστρία το 14% των ανθρώπων ε, κινδυνεύουν ε, ε, από φτώχεια το οποίο σημαίνει ότι το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το 60% της μέσης, του, μέσου εισοδήματος και για τους μερικώς απασχολούμενους το ποσοστό αυτό είναι 11% ενώ για τους άνεργους είναι 38% το οποίο σημαίνει ότι η μερική απασχόληση μειώνει τον κίνδυνο και δεν τον αυξάνει. Και σε ευρωπαϊκές μελέτες ε, βλέπουμε τέτοια στοιχεία. Έχω δει τα ποσοστά ε, από τη ε, μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δείχνουν ότι η φτώχεια όταν, στους εργαζομένους συνήθως έχει να κάνει με, όχι τόσο πολύ με τις άτυπες μορφές απασχόλησης, αλλά με την ελάχιστη δουλειά. Και φαίνεται ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αύξηση του κινδύνου για φτώχεια ε, στους εργαζομένους. Εμένα αυτό με εξέπληξε κάπως, αλλά το βρήκα αυτό στην μελέτη. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι, ε, για παράδειγμα, του ΟΣΑ που δείχνουν ε, ποιοι παράγοντες οδηγούν σε φτώχεια. Και βλέπουμε εδώ μεγάλο ποσοστό ε, ιδιωτικών παραγόντων. Οι προβληματικές ε, μορφές απασχόλησης ε, δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να είναι προβληματικές οι άτυπες μορφές απασχόλησης, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για φτώχεια, αλλά θα πρέπει να εξετάσει κανείς προσεκτικά, και, διότι συχνά είναι άλλοι παράγοντες πιο σημαντικοί η ανεργία και οι ιδιωτικές περιστάσεις ε, είναι πιο σημαντικοί παράγοντες. Ακούσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αυστρία η μερική απασχόληση από τις άτυπες μορφές ε, απασχόλησης είναι ε, η πιο επικίνδυνη. Αλλά τολμώ να πω ότι στην, Γερμανία, στην Αυστρία συγγνώμη, δεν οδηγεί σε επισφάλεια ή μερική απασχόληση. Ε, όσον αφορά τις ε, συμβάσεις μερικούς απασχόλησης αορίστου χρόνου, είναι ελάχιστος ο κίνδυνος επισφάλειας. Ε, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο γιατί είναι ακούσια μερική απασχόληση και εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε πόσο συχνά η μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκούσια και πόσο συχνά είναι ακούσια. Ε, η Eurostat ε, έχει πολύ καλά δεδομένα πάνω στο θέμα αυτό. Εδώ βλέπετε το ποσοστό των ακουσίως μερικώς απασχολούμενων. Αριστερά είναι χαμηλά τα ποσοστά, δεξιά όμως βλέπουμε ότι πάνω από το 70% των ε, μερικώς απασχολούμενων στην, Ευρώπη θα στην Ελλάδα θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο. Ακολουθεί η Κύπρος και η Ισπανία, ενώ βλέπουμε πολύ χαμηλά ποσοστά στην Τσεχία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, τις κάτω χώρες, τη Γερμανία κλπ. Εδώ τι μας κάνει εντύπωση, ότι στις χώρες με υψηλή ανεργία υπάρχει και υψηλό ποσοστό ακούσιας ε, μερικής απασχόλησης. Ενώ σε χώρες με χαμηλή, χαμηλά ποσοστά ανεργίας, ε, οι περισσότεροι μερικώς απασχολούμενοι εργάζονται εκουσίως ε, μόνο με μερική απασχόληση. Θα μπορούσαν δηλαδή να βρουν απασχόληση, πλήρη απασχόληση, δεν το επιθυμούν όμως για κάποιους λόγους. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω κάποιες ε, πτυχές που αφορούν την ε, Αυστρία. Ε, έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ευρώπη μετά τις κάτω χώρες και στους άντρες αλλά κυρίως στις γυναίκες. Ποιο... Ποιες είναι οι αιτίες και ποιο είναι το αποτέλεσμα έχει αυξηθεί πολύ το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Αυστρία. Και ο μέσος χρόνος απασχόλησης ε, πέφτει κάθε χρόνο κατά ένα τέταρτο της ώρας ανά εβδομάδα. Διότι αυξάνεται ο αριθμό των μερικών απασχολούμενων. Βλέπουμε δηλαδή μείωση του χρόνου εργασίας ε, στην Αυστρία. Αυτό πιστεύουμε ότι ανακουφίζει σε κάποιο βαθμό τι ε, αγορέ εργασίε ε, και μπορεί να σας ε, εκπλήσει ότι εκπρόσωπος των εργοδοτών λέει κάτι θετικό ε, σχετικά με την μείωση του χρόνου εργασίας. Ε, εδώ όμως δεν πρόκειται για νομοθετημένη μείωση των ωρών εργασίας όπως είδαμε στη Γαλλία. Στην Αυστρία έχουμε μεγάλη ζήτηση για τη μερική απασχόληση. Το 87% των μερικών απασχολούμενων εργάζονται εκουσίως στην περινή στη μερική απασχόληση. Ε, ένας λόγος ε, για αυτό είναι οι συνθήκες πλαίσιο, διότι οι μερικώς απασχολούμενοι δεν πληρώνουν φόρο ε, δεν πληρώνουν κοινωνικά ασφάλιστρα και επίσης υπάρχουν επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης. Επίσης, ε, χάνει κανείς ε, τα κοινωνικά επιδόματα μόνο από ένα κατόφλι και πάνω. Δηλαδή, αν ε, περάσω από τη μερική απασχόληση στην πλήρη απασχόληση, έχω δύο μειονεκτήματα. Θα πρέπει να πληρώσω φόρο εισοδήματος και χάνω και, τις, και τα κοινωνικά μου επιδόματα. Δηλαδή, η μερική απασχόληση είναι ελκυστική στην Αυστρία και ειδικά για τις γυναίκες μπορεί να είναι μια πολύ γλυκιά παγίδα και όχι ο εργοδότης συχνά συχνά, αλλά ο εργαζόμενος ή μάλλον η εργαζόμενη έχει πολύ λίγα κίνητρα για να περάσει στην πλήρη απασχόληση. Με αυτά θέλω να πω ότι οι άτυπες μορφές απασχόλησης ε, συχνά επιλέγονται εκουσίως και δεν επιβάλλονται από τον εργοδότη ή από άλλους. θα ξεπεράσω αυτήν την ε, διαφάνεια έχει να κάνει με την οριακή μερική απασχόληση στην Αυστρία, όπου έχουμε μεγάλη αύξηση. Η πολύ χαμηλή μερική απασχόληση ε, μπορεί να είναι πολύ ελκυστική όσον αφορά τις συνθήκες σε πλαίσιο ε, κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μερική απασχόληση που δεν ανέφερα ε, είναι ε, οι δυνατότητες φροντίδας των παιδιών και στην Αυστρία συχνά οι παιδικοί σταθμοί για παράδειγμα κλείνουν μεσημέρι οπότε οι γυναίκες θέλουν μερική απασχόληση. Επανέρχομαι λοιπόν στην οριακή μερική απασχόληση. Ήδη στη μερική απασχόληση αλλά και στην οριακή μερική απασχόληση βλέπουμε ε, υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Είναι ελκυστική, ε, συχνά όμως πετυχαίνει ε, το αντίθετο από τον στόχο, δηλαδή πολλές γυναίκες παραμένουν στη μερική απασχόληση αντί να περάσουν στην πλήρη απασχόληση. Επίσης, όσον αφορά την κοινωνική προστασία των άτυπων μορφών απασχόλησης στην Αυστρία, ε, όλες οι μορφές απασχόλησης στην Αυστρία ε, υποχρεωτικά πρέπει να παρέχουν ασφάλιση. Αυτό ισχύει και για τους ε, αυτοαπασχολούμενους. Μάλιστα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας αν ήταν πριν υπάλληλοι. και όσον αφορά την ε, ασφάλιση υγείας ε, είναι ίσες οι προϋποθέσεις για ε, ελεύθερους επαγγελματίες και για υπαλλήλους. αλλά το εργασιακό δίκαιο, οι συλλογικές συμβάσεις και οι ελάχιστοι μισθοί ισχύουν μόνο για τους υπαλλήλους. Επίσης ε, δεν επιτρέπονται οι συμβάσει μηδενικού χρόνου στην Αυστρία, αυτό το έχουν απαγορεύσει τα δικαστήρια. Γενικά το ε, σύστημα της Αυστρίας ακολουθεί την αρχή του flex security. Ε, νομίζω ότι είναι ε, πολύ επίκαιρο το σύστημα αυτό, διότι με ισχυρή κοινωνική προστασία οδηγεί σε ευελιξία το σύστημα αυτό, το οποίο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ε, γενικά ε, είναι, οι αυτοαπασχολούμενοι γενικά είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη θέση τους. Επίσης, ε, όσον αφορά τις άτυπες μορφές απασχόλησης και την αγορά εργασίας, είναι σαφές ότι και εδώ υπάρχει μια ισορροπία. Έχουμε δει πολύ πιο σημαντικές διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας ε, από την νωρίτερα. Γι' αυτό θέλουμε ευελιξία. και εάν οι εργοδότες ε, δεν ε, το πετυχαίνουν ε, αυτό, τότε ζητούν προσωρινές συμβάσεις. Εάν όμως έχω την ευελιξία, τότε δεν έχω κίνητρα για να επιλέξω άλλες μορφές απασχόλησης. Ο πρόεδρος ε, του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο κύριος ε, Σμιτ, λέει ότι οι βάσει ε, του γερμανικού οικονομικού θαύματο ήταν οι ευέλικτε μορφέ απασχόλησης και ο καθορισμός των μισθών. Και Υπουργό Απασχόλησης και Οικονομικών της Γερμανίας, ο Βολφκαν Κλέμεντ, πρώην είπε ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να φέρουμε τους ανθρώπους στην απασχόληση από την προσωρινή απασχόληση. Εάν θέλει κανείς να ρυθμίσει τις άτυπες μορφές απασχόλησης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πολλοί από τους ανθρώπους ότι πολλές μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι άτυπες μορφές απασχόλησης ε, έχουν θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, ε, ότι ιδιαίτερα για ε, ανθρώπους ε, ανέργους για πολύ καιρό είναι ελκυστικές αυτές οι θέσεις απασχόλησης και αν δεν καταφέρω να δημιουργήσω αρκετές θέσεις απασχόλησης, μάλλον αν καταφέρω να δημιουργήσω αρκετές θέσεις απασχόλησης, οι άτυπες μορφές εργασίας θα εξαφανιστούν από μόνες τους. Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην ε, ευελιξία στις μόνιμες θέσεις απασχόλησης ε, και την ε, ελκυστικότητα στις άτυπες μορφές απασχόλησης. Το flexicurity συνεχίζει να είναι επίκαιρο, δηλαδή ο συνδυασμός ισχυρής κοινωνικής προστασίας και φιλελεύθερων μορφών απασχόλησης. Ε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ε, έχουμε, πολλές, ε, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις συνθήκες εργασίας και γι' αυτό είναι λογικό να υπάρχουν και πολύ διαφορετικές μορφές απασχόλησης σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκλάισνερ. Η παρουσίασή σας μας έδωσε μια σαφή εικόνα με στοιχεία και μας δείχνει και την πολύ, καλή πολύ καλή κατάσταση στην Αυστρία. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζει ε, την κατάσταση σε άλλα μέρη της Ευρώπης όπου μπορεί να υπάρχει υψηλή ανεργία. Και όπως λέω εγώ πάντα, αν δεν υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι που να επηρεάζουν ε, την πολιτική στην αγορά εργασίας σε μια χώρα, τότε αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εάν όμως υπάρχει αυτό, τότε μπορούμε να έχουμε μια πολύ θετική εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ε, λόγο τον δίνω στον συνάδελφό μου, ε, Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σιλικιώτη, που είναι και η συγητής ε, της σχετικής έκθεσης. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. I will speak in Greek, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου για την πρόσκληση να τοποθετηθώ σε μια ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση. Επιτρέψτε να πω πως τέτοιες εκδηλώσεις ενδυναμώνουν την τάση που καταγράφεται εδώ στο Κοινοβούλιο το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα ότι δεν μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στην επισφάλεια στην οποία οδηγούνται. Είναι όντως καιρό να γνωριστεί πως η καταστροφή του κοινωνικού κράτους, η πίεση πάνω στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Απειλούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και έδωσαν, αν θέλετε, την αφορμή για την αύξηση των μη τυπικών συμβολέων και άτυπων μορφών απασχόλησης και εν τη της απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων. Το δικό μου επιχείρημα είναι πως η αύξηση των μη τυπικών συμβολέων εργασίας φτωχοποιεί τους εργαζόμενους και δεν αποτελεί τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας. Ε, και φάνηκε αυτό και από τις έρευνες. Ε, η σημερινή φαινομενική αύξηση των ποσοστών απασχόλησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβει σε πολλές περιπτώσεις την αύξηση των συμβολέων μηδενικών όρων τη ψευδή αυτοαπασχόληση και θέση εργασίας με ακούσια συμβόλαια μερική απασχόλησης, οι οποίε δεν παρέχουν αξιοπρεπή ζωή και όλα τα εργασιακά δικαιώματα στους εργαζομένου. Η αντίδραση όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το πρόβλημα. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται αλλαγή πλεύση. Στο τέλο τη παρέμβαση μου θα θέσω κάποιε εισηγήσει για προβληματισμό, οι οποίε εν μέρει καταγράφηκαν και στην έκθεση με τίτλο Συνθήκε εργασία και επισαφαλή απασχόληση, στην οποία ήμουν εισηγητή. Οι πλήστοι των σημερινών ομιλητών έδωσαν παραδείγματα τη αύξηση τη επισφάλεια στην απασχόληση. Και συμφωνώ με αρκετά από τα συμπεράσματα. Από τη στιγμή που το δίχτυ κοινωνική προστασία των εργαζομένων αφαιρείται, η διαπραγματευτική ικανότητα των εργαζομένων μειώνεται. Το αποτέλεσμα, πολλοί εργαζόμενοι να αναγκάζονται να αποδέχονται συμβόλαια με χαμηλότερους μισθούς, με λιγότερα δικαιώματα και με περιορισμένη διάρκεια. Επίσης, είναι πλέον ξεκάθαρο πως τα μη τυπικά συμβόλαια εργασίας και τα συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας δεν είχαν πραγματικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της ανεργίας και την αποτελεσματική μείωση των ποσοστών τη. Αυτό αποδεικνύεται και μέσα από άλλες ερευνές που έγιναν εκ μέρους των οργάνων και στουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όμως η έρευνα που έγινε εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης αυτού του Κοινοβουλίου αναφορικά με την επισφάλεια στην εργασία δείχνει ξεκάθαρα πως οι εργαζόμενοι με συχνά επιβεβλημένα συμβόλαια περιορισμένη διάρκεια και μερική απασχόληση αυξήθηκαν σημαντικά στην Ένωση τα τελευταία 15 χρόνια. Η τυπική απασχόληση δηλαδή τα, ε, η, τα συμβόλαια ορίστου χρόνου, μειώθηκαν από 62% το 2004 στο 59% σε 10 χρόνια. Τέσσερις στους 10 εργαζόμενους εργάζονται πλέον μόνιμα με συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας, ενώ περίπου 4% των εργαζομένων παραδέχονται πως δούλεψαν σε αδήλωτη εργασία τους τελευταίους 12 μήνες. Μπορεί τα συμβόλαια αυτά να υπήρχαν και πριν την οικονομική κρίση, Εν τούτης, οι ανεπαρκείς και κοινωνικά κατάλληλες λύσεις που δόθηκαν για καταπολέμηση της κρίσης όξυναν την επισφάλεια στην εργασία. Τέτοιες ακατάλληλες λύσεις ήταν οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν σε διάλυση του κοινωνικού ιστού και τη φτωχοποίηση μεγάλων τιμάτων του πληθυσμού, κυρίως των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Σε τελευταία του έρευνα, το Ινστιτούτο Eurofound έδειξε τη σχέση μεταξύ των εργασιακών πολιτικών και τη στόχια στην εργασία. Σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση αυξήθηκε ο κίνδυνο τη στόχια στην εργασία και η ηλική στέρηση, η στέρηση αγαθό. Ενώ τα μόνιμα συμβόλαια μειώνονται, ο κίνδυνο στόχια των εργαζομένων με συμβόλαια περιορισμένη διάρκεια ανέβηκε στο 15%. Μια κοινωνική ομάδα που δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα ήταν νέοι. Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, περίπου 4 με 6 εκατομμύρια νέοι το χρόνο απασχολούνται σε πρακτικές ασκήσεις. Αυτό μας δείχνει ένα ανησυχητικό φαινόμενο, αν σκεφτεί κάποιο πως οι πλήστε αυτών των ασκήσεων συνήθως δεν παρέχουν εργασιακά δικαιώματα στους νέους και πολλές από αυτές είναι μάλιστα και απλήρωτες. Επίσης, παρόλο που σύμφωνα με την έρευνα των 90% των νέων που συμμετέχουν σε πρακτική εξάσκηση θεωρούν την άσκηση του αυτή πολύ βιοθητική, εν η άσκηση αυτή δεν τους οδηγά σε θέση εργασίας. Κατά συνέπεια, αυτό το σύστημα λειτουργεί εν μέρει αντιπαραγωγικά. Αντί οι νέοι να πληρώνονται αξιοπροπώς για τη δουλειά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματα ενός εργαζομένου, γίνονται μοχλός πίεσης από τους εργοδότες προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ο κίνδυνος που νομίζω βγαίνει από την ίδια την έρευνα είναι πως οι νέοι άνθρωποι γίνονται σε πολλές περιπτώσεις προϊόν εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα όταν το κράτος δεν βάζει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο στις πρακτικές ασκήσεις εργασίας. Την ίδια ώρα και πάλι η έρευνα του Eurofound παρουσιάζει τις μορφές εργασίας στις οποίες γίνεται περισσότερη κατάχρηση και χρησιμοποιούνται παράνομα. Το Eurofound συνόψισε το δικό του ορισμό στα δύο χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει η απάτη ή ε, fraudulent ε, στην εργοδότηση. Πρώτο είναι η υπερολαβία κάτω από τη μορφή άλλου συμβολέου και δεύτερον οι συνθήκε απασχόληση ενό εργαζομένου δεν ανταποκρίνονται στου επίσημου όρου του συμβολέου του. Τα κύρια αποτελέσματα είναι πω οι κύριε μορφέ απασχόληση που παρουσιάζουν αύξηση στι μορφέ απάτη, είναι αυτοαπασχόληση περίπου 23,5% συμβόλαια περιορισμένη διάρκεια περίπου 16%, απόσπαση εργαζομένων 15%, προσωρινή εργασία περίπου 13%, Πρακτικέ ασκήσει 11%, Υπεργολαβίε μέσα στην ίδια την εταιρεία ή μεταξύ εταιρείων 10%, on-call και εποχιακή εργασία 7%. Τα πιο πάνω δείχνουν πόσο επικίνδυνη ήταν η απορρίθμιση της εργασίας πριν και κατά την οικονομική κρίση. Δυστυχώ όμω η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εντελώ αποθαρρυντική. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων για τον κοινωνικό πυλώνα μεταξύ των αρχικών των κρατών στο Κέντεμποκ, που αναφέρθηκε προηγουμένω η αγαπητή συνάδελφο και πρόεδρο τη Επιτροπή, η Σίλια Ουίστρο, απόδειξαν πω ο πυλώνα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κοινωνικό πλασέμπο. Ένα προπέτασμα καπνού όπως εύστοχα το χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός τύπος. Δεν υπάρχει καμιά νομική δέσμευση προς τα κράτη-μέλη, κάτι που σίγουρα δεν επιτρέπει στον κοινωνικό πυλώνα να γίνει πραγματικά πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο του είναι πολύ γενικό και μιλά ξεκάθαρα για την αναγκαία ανευελιξία των εργοδοτών. Ούτε λέξη όμως για το ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία. Αντίθετα, η Κομισιόν προωθεί παράλληλα μέτρα προ την κατεύθυνση τη περαιτέρω φιλελευθερωποίηση και τη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Την ίδια στιγμή που καλεί του κοινωνικού εταίρου για συζήτηση, προωθεί τα μέτρα όπω η καταπολέμηση τη γραφειοκρατία εισαγωγικά στον τομέα τη εργασιακή ασφάλιση. Αγαπητοί φίλοι, από τα πιο πάνω δεν μπορεί να εξαχθεί άλλο συμπέρασμα από ότι τα μη τυπικά συμβόλαια εργασία δυστυχώ δεν μπορούν να δώσουν λύσει στην αργία. Αντίθετα στι πλήστε φορέ οδηγού στη φτωχοποίηση και την κοινωνική ενέργεια. Την ίδια δώρα ο κοινωνικό πυλώνα αποδείχτηκε απλό προπέτασμα καπνού και δεν προβλέπεται αλλαγή πλεύση από τα κράτη-μέλη. Έτσι η εργοδοτική πλευρά μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητη με την προσφορά άτυπων και επισφαλώς συμβολών απασχόληση ε, όταν δεν προσφέρεται ακόμα και παράνομα συμβόλαια. Η λύση στο πολύπλοκο αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να περιοριστεί δημιουργία νέων παρενώσεων προς τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται άμεσα μια αλλαγή πλεύσης από τις πολιτικές της ανεξέλεκτης αγοράς και της λιτότητας. Εμείς, μέσα από την έκθεση που ετοιμάσαμε στο Κοινοβούλιο, προτείναμε την επαναφορά της έννοιας της απασχόλησης σωστή της βάση. Η απασχόληση πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να προσφέρει στον εργαζόμενο και την οικογένεια του μια ισορροπημένη ζωή. Στην έκθεση μα, που υπερψηφίστηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, καταφέραμε μαζί με του κοιόδη ηγητέ να κάνουμε βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο του ILO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, για την αξιοπρεπή απασχόληση που ορίζει την αξιοπρεπή εργασία ω πλήρη και παραγωγική απασχόληση που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, ένα δίκαιο εισόδημα και ασφάλεια στην εργασία που παρέχει ελευθερία της έκφρασης της άποψης, της οργάνωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές τους και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση για όλους άντρες και γυναίκες. Για να επιτευχθεί αυτό, το πρώτο βήμα πρέπει να κάνει, που πρέπει να κάνει η Ένωση είναι να προωθήσει πολιτικές που θα ενδυναμώσουν τους εργαζόμενους μέσω του κοινωνικού διαλόγου και της επέκτασης το συλλογικό διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντα πω όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμα τη συνάθρηση και τη συλλογική διαπραγμάτευση ελεύθερα και χωρί φόβο. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν στρατηγικέ καθολική κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικέ συμβάσει και κατοχύρωση του ρόλου των συνδικάτων ω κοινωνικών εταίρων να καταδικαστούν οι καταχρήσει που γίνονται στα πλαίσια πρακτικών ασκήσεων ή ευέλικτων συμβολών εργασία. Υπενθυμίζομαι πω σύμφωνα με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε εργαζόμενο έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστη διάρκεια εργασία, σε ημερήσιε και εβδομαδιαίε περιόδου ανάπαυση, καθώ και σε αιτήσια περίοδο αμοιβαίνων διακοπών. Την ίδια ώρα προφανώ χρειάζεται δυνάμωση του κοινωνικού κράτους αλλά και πολιτικές δημιουργίας αξιοπρεπό θέσεων. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο δυναμώνουν οι φωνές για πραγματική εισαγωγή του δικαιώματος της αξιοπρεπής εργασίας στην εθνική αλλά και ενωσιακή νομοθεσία. Συνεπώς, ως δεύτερο βήμα προτείνομαι ναι. Ε, την εισαγωγή μιας οδηγίας πλαίσιο για την πρόθεση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τις μορφές απασχόλησης, διασφαλίζοντας για κάθε εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων. Τρίτον, υποστηρίζουμε την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να δοθούν τα εργαλεία για αλλαγή των πιο αντεργατικών τυχών της ε, ενιαία αγορά και του πλαισίου οικονομική ε, διακυβέρνηση. Και τέλο, αυτό που απαιτείται είναι τροποποίηση το συνθήκων ώστε να εισαχθεί ένα πρωτόκολλο κοινωνική πρόοδου το οποίο έμπρακτα να θέτει τα κοινωνικά δικαιώματα πάνω από τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση ε, της Επιτροπής Απασχόλησης ε, ε και την άποψή σα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την επισφαλή εργασία στην Ευρώπη. Ο κύριο Μπέκερ δυστυχώ έπρεπε να αποχωρήσει. Ε, θα συντονίσω λοιπόν λίγο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Να σας συστηθώ, θα σα συστηθώ μάλλον εντό ολίγου. Ε, προς το παρόν είμαι η Τζουν Κίρτον Ντάρλινγκ, ε, σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πλήρε μέλο ε, τη επιτροπή Αναφορών. Έχουμε περίπου ένα τέταρτο για ερωτήσει και απαντήσει. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ζητήσω ρωτήσω από τους συναδέλφους εδώ στην αίθουσα, αν θέλουν το λόγο. Έχουμε ένα πρώτο μιλητή. Ξεκινάμε λοιπόν. Σας παρακαλώ να είναι σύντομες οι ερωτήσεις για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να λάβουμε και αντίστοιχα σύντομες απαντήσεις. Ο κύριος Βαλέσα. Τρεις ερωτήσεις έχω για τη χώρα μου κυρίως. Υπάρχουν ε, νομοθετικές αλλαγές οι οποίες να οδήγησαν σε αυξανόμενο μερίδιο προσωρινής απασχόλησης όπως για παράδειγμα στην Ισπανία η αύξηση της προσωρινής απασχόλησης είναι χαρακτηριστική για την Πολωνία ή έχουν αντίστοιχες τάσεις και άλλες χώρες. Και τέλος, ε, ποιοι είναι οι παράγοντες ε, που καθορίζουν σε νομοθετικό επίπεδο το μεγάλο μερίδιο της προσωρινής ε, και άτυπης απασχόλησης και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελεόνα Ευχαριστώ, Τζουν. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρεμβάσεις. Ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο και λεπτό πραγματικά. Είναι μεγάλη μάστιγα η επισφαλής εργασία στην Ευρώπη και στην Ιταλία. Εγώ σκέφτομαι και τη χώρα μου. Ε, εγώ ε, όμως θεωρώ ότι μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό φέρουν και οι θεσμικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια απέφυγαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ε, για να ξαναδώσουν αξιοπρέπεια στους εργαζομένους και να τους ε, ε, ε, δώσουν τα δικαιώματά τους. Είναι πολύ ευρύ το πρόβλημα, δεν μπορεί να πρόκειται για απλή αμέλεια. Εγώ διαβλέπω πραγματικά ε, διάθεση να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς του χώρου της εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας για να επιβάλλουμε την κυριαρχία της ανταγωνιστικότητας χωρίς κανένα δισταγμό. Και ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε η εργασία να είναι μέσω αξιοπρέπειας. Εγώ θεωρώ και θα ήθελα και εδώ και την άποψή σας ότι υπάρχει μεγάλη ε, υποχώρηση από πλευράς ε, νομοθέτη, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη, με μοναφικό στόχο αυτή την ε, τόσο συχνά επικαλούμενη ευελιξία που θέλει να χρησιμοποιηθεί ως ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να καταστρέψουμε και να μειώσουμε την προστασία που προβλέπεται στην εργασία. Και όλο αυτό καταπατώντας και αγνοώντας πλήρως τις ε, πάρα πολλέ καταγγελίε που έχουν γίνει ε, σύν το χρόνο και από αναφέροντε εδώ στην Επιτροπή μα, για παράδειγμα. Ε, και υπήρχαν ένα σωρό προβληματισμοί διακρίσεις ε, μεταξύ εργαζομένων με συμβάσει αορίστου και ορισμένου χρόνου και το καθεξής. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι πολύ σύντομη και θα πάω στο προκείμενο. Η ερώτηση αφορά την ε, εξαιρετική ε, νομοθεσία την 1999-70. Μήπως θεωρείτε ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αυτή η οδηγία ίσως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επί τη βάση ποιων νομικών υποδείξεων ακριβώς για να αποφύγουμε αυτή η ευελιξία να μην συνεχίσει να είναι ευφυή εφιάλτης για τους εργαζομένους που εργάζονται με αυτές τις επισφαλείς ε, ζωφερές συνθήκε. Ευχαριστώ κυρία Βαλένα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να επενθυμίσω κάποια στοιχεία της Eurostat αυξήθηκαν οι φτωχοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1 εκατομμύριο 700.000 παρά το γεγονός ότι ο στόχος της Ευρώπης 2020 είναι να έχουμε 20 ε, εκατομμύρια ε, λιγότερους ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας μέχρι το 2020. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα ήθελα να δω αν μου πείτε τα στοιχεία αν γνωρίζετε. Θα ήθελα να ξέρω πόσα ήταν τα επισφαλή συμβόλαια που έγιναν στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης και επίσης ποιος ήταν ο ε, καθαρός αριθμός ε, επισφαλούς εργασίας που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 και μετά. Και αν περάσουμε τώρα στο θέμα των γυναικών, ε, βρίσκονται 10 μονάδες ε, κάτω από το ποσοστό της απασχόλησης ε, και ε, αν μιλήσουμε και για τις γυναίκες της υπαίθρου και τη δουλειά τους η οποία είναι αόρατη, τι γίνεται με την επισφαλή εργασία στην υπαίθρο για τις γυναίκες. Και θα ήθελα να πω ότι στην ΕΣΠΙΑ υπάρχουν κάποιες συμβάσεις οι οποίες ε, ε, είναι πονίδιστο, αλλά είναι ακόμα και συμβάσεις μίας ώρας. Ε, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει μετά από τον πόλεμο στην Ισπανία. Δηλαδή η φιγούρα του φτωχού εργανοζομένου, που ούτε καν με δύο θέσεις εργασίας δεν μπορεί στο τέλος του μήνα να καλύψει τα έξοδα της οικογένειάς του και της διαβίωσής του. Και θα ήθελα να κάνω και συγκεκριμένη ερώτηση στον συνάδελφο τον Νεοκλή, ο οποίος ήταν και εισηγητής για την έκθεση και θα ήθελα να το συγχαρώ γιατί το αρχικό σχέδιο έκθεσης ήταν πάρα πολύ εύρωστο και λέγε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να την χάνουν κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να μου εξηγήσει τι συνέβη στο μεταξύ ε, με, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των τροπολογιών και εξαφανίστηκαν όλα Όλε αυτές οι ρητές αναφορές. Τι πρόβλημα διαπιστώθηκε κατά τη διαπραγμάτευση και την ψηφοφορία της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Εντουάρ. Ναι, ευχαριστώ. Κάποιες παρατηρήσεις ε, πριν ε, κάνω ερωτήσεις. Ο κύριος ε, Γκλίσνερ μας μίλησε για την κατάσταση στην Αυστρία. Άκουσα βέβαια το τέλος της παρουσίασής του μόνο και ζητώ συγγνώμη. Ε, τι ζούμε στην πραγματικότητα στην Ευρώπη όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και την πολιτική της απασχόλησης. Όλα αυτά ξεκίνησαν ε, από τη Γερμανία και από εκεί και πέρα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, ακολούθησαν τη Γερμανία και τώρα έχουμε κάνει το γύρο των 28 διότι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πρέπει εντός εισαγωγικών και βάζω πολλά εισαγωγικά εδώ να εξυγχρονίσουμε την αγορά εργασία. Εξυγχρονισμό σημαίνει ευελιξία, επισφάλεια πάνω απ' όλα. Και πριν έρθω εδώ μιλούσαμε για την κατάσταση των Ισπανών εργαζομένων. Το 20% το φτωχότερο είναι αυτοί οι οποίοι βίωσαν πλήρω τι συνέπειε της κρίσης και δεν ξέρω, δεν το άκουσα στην αρχή, μπορεί να το είπατε και στην αρχή, υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι ε, μερικής απασχόλησης που μπορεί να είναι εξαιρετικό παράδειγμα σε κάποιες χώρες, αναφέρομαι στην Ισπανία αλλά και στην Γαλλία, κάποιες φορές επιβάλλεται αυτή η μερική απασχόληση. Διότι ο νόμος προβλέπει, και εδώ απαντώ και στη, σχολή, ε, συνάδελφο και θα συμφωνήσω μαζί της, αν πάρετε δύο θέσεις ε, μερικής απασχόλησης, δεν αμείβεστε σαν να είχατε μία ε, μόνιμη θέση απασχόληση. Στην Ισπανία, στον τομέα των υπηρεσιών, είμαστε μεταξύ 20 και 33% μείωση των ε, μισθών. Όχι κερδίζουμε παραπάνω, αλλά μειώθηκαν οι μισθοί κατά 20 με 33%. Αυτό ισχύει και για τον κλάδο του τουρισμού και για τον κατασκευαστικό κλάδο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πάρα πολύ φιλελεύθερη κατάσταση, όπου πραγματικά ε, το κόστος για τις χώρες περνάει από το εργατικό δυναμικό, πρέπει να είναι ευέλικτο και πρέπει να είναι και φθηνό. Και πολλέ χώρε μα ε, τίνουν, το λέει και η Γαλλία για παράδειγμα η χώρα μου, ότι κοιτάξτε τι κάνουν στην Ισπανία, λειτουργεί. Ε, το 80% των συμβάσεων είναι συμβάσει λιγότερο του ενό μήνα. Αυτό το μοντέλο θέλουμε. Και εδώ βλέπουμε και τα σφάλματά μα και τι αδυναμίε μα. Η κοινωνική πολιτική δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι καν ε, επιμερισμένη αρμοδιότητα. Πρέπει πραγματικά λοιπόν να δούμε τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τα θέματα αυτά. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δω είναι πέραν του να πούμε τι ωραία που πηγαίνει το μοντέλο της Αυστρίας, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι ο αντίκτυπος και για την ανάπτυξη και για την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Αυστρία. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω και ένα σχόλιο από πλευράς μου για αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ευρώπη για τα δυστεόρατα ύψη της ανισότητας που έχει συνέπειες και για την κοινωνική συνοχή και τε, άμεσες και συνέπειες για την ε, εμπιστοσύνη στα, ε, ε, στους δημόσιους θεσμούς, στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και στο ευρωπαϊκό όραμα, που για μένα αυτό είναι κομβικό ερώτημα που κανένας από εσά δεν έθεσε. Είναι και σημαντικό από οικονομική σκοπιά, αλλά υπάρχει και μια πολιτική διάσταση στην επισφάλεια της εργασίας, διότι μπορεί να δημιουργήσει ε, και το σπόρο για πάρα πολύ επικίνδυνες ε, πολιτικές κινήσεις ε, και πολιτικές αλλαγές και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα αυτής της συζήτησης. Έχουμε λίγο χρόνο, θα κλέψω και λίγο χρόνο από το επόμενο πάνελ. Προεδρεύω εγώ, μπορώ να κάνω τι θέλω. Δεν θα κάνω μακρά εισαγωγή για την υποφαινόμενη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να σας δώσω ολονών Α, συγγνώμη, ένα ακόμα σχόλιο πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομο. Η κυρία Κούνεβα. Σύντομη, μόνο ένα λεπτό αν γίνεται. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω το, Euro, το Eurofound αν μπορούν να μας πούν γιατί το 78% των Ελλήνων δουλεύουν ακουσίως στη μερική απασχόληση λόγω μισθών ή συνθηκών εργασίας και τι άλλα ευρήματα έχουν από αυτό το θέμα ε, για, το Ευρωπαϊκό Νότο. Σα Σας ευχαριστώ. Θα κλέψουμε λοιπόν λίγο χρόνο από το επόμενο πάνελ. Παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Θα είμαι πολύ αυστηρή ε, με το σφυράκι μου εδώ πέρα, αν σημαδεύσω σωστά. Ε, κύριε Μπιλέτα... 1,5 λεπτό αν είναι δυνατόν για να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ε, και τον ίδιο χρόνο θα δώσω και στους άλλους. Ξέρω ότι είναι πολύ λίγος χρόνος. Να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση. Δεν έχω στοιχεία, δεν ξέρω τα στοιχεία απ' έξω, θα το εξετάσω όμως και θα στείλουμε τα στοιχεία στην ε, κυρία Ευρωβουλευτή. Νομίζω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις ε, απευθύνονταν ε, σε κάποιους από τους άλλους ομιλητές. Αν θέλετε να επανέλθω μετά τους άλλους. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσω να σας δώσω κι άλλο χρόνο, αλλά εκτιμώ την αλληλεγγύη σας που δίνετε περισσότερο χρόνο ομιλία στους άλλους ομιλητές. Ε, η κυρία Μάκτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να απαντήσω στις ερωτήσεις μία προς μία. Δεν υπήρξαν ε, νομοθετικές αλλαγές στο πολωνικό πλαίσιο που να οδηγήσουν σε αύξηση της ε, μερικής απασχόλησης. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι είδαμε μια ε, βαθμιαία αύξηση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε τον ρόλο του δημοσίου τομέα που υπονόμευσε τα πρότυπα στην απασχόληση, διότι υπήρξαν αρκετέ ε, περιπτώσει εξωτερικής ανάθεσης ε, στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή. Και οι ε, εργαζόμενοι που έχασαν καλές θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο τομέα προσλήφθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες όμως εργάζονταν με βάση ε, διαγωνισμούς ε, με μόνο παράγοντα το, τη χαμηλή τιμή και έτσι κατέληξαν σε πολύ κακέ ε, θέσεις απασχόλησης στην Πολωνία. Συχνά θεωρούμε ότι αυτό είναι πολωνικό φαινόμενο, αυτές οι κακές ε, συμβάσεις εργασίας ε, και οι συμβάσεις μηδενικού χρόνου, αλλά από ό,τι ακούμε εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καθαρά ε, πολωνικό φαινόμενο. Η φύση αυτών που βλέπουμε είναι παρόμοια σε ίσως όχι όλα τα κράτη-μέλη, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιοι μπορεί να είναι οι νομοθετικοί παράγοντες ε, ε, της επισφάλειας ε, και της προσωρινής απασχόλησης. Ακούσαμε πολλά στην έκθεση που παρουσιάστηκε, νομίζω όμως και ως οικονομολόγος μιλώ, τίθεται το θέμα του κόστους πρόσληψης και απόλυσης. Αν υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί αυτό το κόστος, γιατί να μην γίνει αυτό. Δεύτερον, και ο φόρος, η φορολογία που συνδέεται με διάφορες μορφές απασχόλησης αποτελεί παράγοντα. Τρίτον, ακούμε πολλά για το franchising, τη δικαιόχρηση ε, οι συμβάσεις ε, ε, περιορισμένου χρόνου κλπ. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν επηρεάσει την κατάσταση στην Πολωνία. Και τέλος, ε, να σας δώσω μερικά στοιχεία. Στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια, ενώ ε, αυξήθηκε ο αριθμός, ε, ο όγκος της απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, είδαμε μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων. Υπάρχει ένα ποσοστό της ε, προσωρινής απασχόλησης, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο ποσοστό, καταφέρει να, να ε, λειτουργήσει ως πέρασμα ανθρώπων από την ανεργία στην πλήρη απασχόληση και να μειώσει τις ανισότητες. Ε, κύριε Κλάισνερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πράγματι, η κατάσταση ε, στην ε, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία διαφέρει πολύ από την κατάσταση σε άλλες χώρες ε, Βέβαια δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει τα δεδομένα ένα προς ένα προς τις, στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. Ωστόσο είμαι πεπισμένος ότι ε, θα πρέπει η επιθυμία μας ε, να είναι οι καλές ε, θέσεις πλήρους απασχόλησης για όλους, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς. Υπάρχει λοιπόν εδώ σύγκρουση στόχων ανάμεσα στις ποιοτικά καλές θέσεις απασχόλησης και τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης μετά την κρίση στην Ευρώπη καθαρά έχουμε ένα πρόβλημα, έχουμε πολύ λίγες θέσεις απασχόλησης και νομίζω ότι είναι καλύτερο το να έχει κανείς άτυπη απασχόληση από το να μην έχει καθόλου. Και αυτή ήταν ε, η βασική ιδέα πίσω από τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, που εφαρμόστηκαν στη Γερμανία και τελικά ήταν επιτυχής ε, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, ε, μείωσαν ε, την ανεργία και μείωσαν την φτώχεια. Γενικά λοιπόν είμαι ικανοποιημένος που φαίνεται ότι η Ευρώπη βγαίνει από την κρίση. Τα τελευταία στοιχεία από την Eurostat δείχνουν ότι η φτώχεια και ο κίνδυνος φτώχειας στην Ευρώπη μειώνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε σχέση ε, εάν συγκρίνουμε παγκοσμίω, ε, είναι πολύ ε, κοινωνικά. Αν συγκρίνουμε δηλαδή με τι Ηνωμένε Πολιτείε, διαπιστώνουμε ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο έχουμε υψηλέ κοινωνικέ δαπάνε, έχουμε και ένα πολύ πυκνό σύστημα ρύθμιση σε σχέση με άλλε χώρε. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει έλλειμμα. Ωραία, σα ευχαριστώ. Ο κύριο Ηλικιώτης. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν να πω ότι η Ευρώπη βγαίνει από την κρίση αυτό δεν αφορά του εργαζόμενου στην μεγάλη του πλειοψηφία. Να απαντήσω στη συνάδελφη την την Βαλίνα ότι υπάρχουν αναφορέ για τι συλλογικέ συμβάσει και την κοινωνική ασφάλιση. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο στο αρχικό κείμενο, ε, λόγω του ότι υπάρχουν συμβιβασμοί για να εγκριθεί μια έκθεση. Είναι σημαντικό όμω ο ορισμό του ΑΕΛΟ. Η δεύτερη μου παρατήρηση, η κρίση κατέδειξε την ασυδοσία τη λεγόμενη ελεύθερης αγοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευελιξία οδηγά στην επισφάλεια. Και επειδή μιλούμε για δεσμευτικούς όρους, δεν μπορεί στην Ευρώπη να έχουμε σύμφωνο σταθερότητας, με οικονομικά κριτήρια δεσμευτικά, να έχουμε περιβαλλοντικά πρότυπα και να μην έχουμε κοινωνικά κριτήρια και δεσμευτικού όρου για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αξιοπρεπή εργασία. Και αυτό πρέπει να είναι η επιδίωξή μα και προ αυτήν την κατεύθυνση σπρώχνει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Θα ήθελα να ολοκληρώσω το ρόλο μου ως κύριος Μπέκερ, ευχαριστώντας το πρώτο πάνελ ε, για όλες τις παρεμβάσεις ε, των ε, ευρωβουλευτών που έλαβαν το λόγο. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ, στο οποίο πλέον είμαι επισήμωση επισήμως η Τζούντ Κερτον Ντάρλινγκ και δεν είμαι ο κύριος Μπέκερ. Και θα ήθελα να σας πω δύο φράσεις ε, για μένα πριν εκλεγώ Ήμουν ε, ερετό μέλος ε, συνδικαλιστικών σωματείων, συμμετείχα στη Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, και είχα επαφές και στην Ευρώπη με τον καλό μου το φίλο τον Εντουάρ, αλλά η εμπειρία μου στον κόσμο των συνδικάτων είναι ότι πολλές φορές η αύξηση της επισφαλούς εργασίας έχει δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις σε αυτούς που βρίσκονται και σε μόνιμες θέσεις εργασίας, συνήθους εργασίας και επιβάλλεται και άτυπη μορφή εργασία σε ανθρώπου που υποτίθεται ότι είχαν μια συνήθι σύμβαση εργασία. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει τόσο μακριά ακόμα στη συζήτηση σε κάποιο βαθμό. Και επίση ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι εκπροσωπώ τη βορειοανατολική Αγγλία. Είναι κατά πάσα πιθανότητα η πιο καλή περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολύ όμορφη. Αλλά έχουμε και την ε, φήμη ότι και φέτος είμαστε η πρωτεύουσα των συμβάσεων μηδενικών ορών της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το καλοκαίρι του 2016 στο 2017 είχαμε αύξηση κατά 30%. 45.000 άνθρωποι στην περιοχή μου, που είναι η μικρότερη περιοχή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, εργάζονται σε πολύ επισφαλείς ε, θέσεις εργασίας, ε, μηδενικών ορών και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο πάνελ ε, όπου θα συζητήσουμε αυτή την προπτική και θα τα δούμε από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων και θα δούμε και την άποψη της Επιτροπής Αναφορών. Έχουμε και κάποιους αναφέροντες που ακούσαμε στο παρελθόν στην Επιτροπή μας οι οποίοι ε, έφεραν αναφορές ε, για την προσωρινή και επισφαλή μορφή εργασίας ε, και ζήτησαν και μέτρα για πρόληψη και επιβολή κυρώσεων για αυτή την κατάχρηση των συμβάσεων ε, αορίστου χρόνου και έχουμε και αυτή την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας αλλά ταυτόχρονα και ασφάλειας για τους εργαζομένους. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, να σας παρουσιάσω το δεύτερο πάνελ. Ο πρώτο ομιλητής θα είναι ο Ιαν Χότσον, ο Εθνικός Πρόεδρος ε, των εργαζομένων ε, σε αρτοπία και ε, στον τομέα της διατροφής, τον Κέρστιν Χάουελ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, Τροφίμων Γεωργίας Τουρισμού Συνδικάτων, τον Βιντσέντσο Ντεμικέλε στη συνέχεια, εμπειρογνώμονα σε σύντομες συμβάσεις εργασίας και νομολογία νομικό και ελέκτρο από την Ιταλία, τον Σέργιο Γκαλεάνο, ζητώ συγγνώμη αν προφέρω λάθος τα ονόματα, είναι εθνική νόσος αυτή, ε, νομικό, ο οποίος εκπροσωπεί Ιταλούς αναφέροντες, ε, το Μάικαλ Άσπρουκ, ε, αναφέροντα ο οποίος εκπροσωπεί συμβασιούχους ε, στο ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τέλος θα ακούσουμε και από τον ε, ε, σημαντικό παράγοντα στην αίθουσα που θέλουμε να ακούσουμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ακούσουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλά από τα σχόλια τα οποία έγιναν και θα γίνουν εδώ σήμερα. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον Ιαν, έχετε 10 λεπτά, ε, μπορείτε ελεύθερα να μην τον εξαντλήσετε το χρόνο σας και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι μηδενικές οι συμβάσεις μηδενικής εργασίας ε, είναι πολύ σημαντικές για συμβάσεις ε, ε, που περιλαμβάνουν ε, ε, όρους που λένε ότι ο εργαζόμενος πληρώνεται μόνο για αυτό για το οποίο δουλεύει, πρέπει να είναι παρόν στη δουλειά και απαγορεύεται να εργαστεί για άλλους εργοδότες παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εργαστεί περισσότερο. Βέβαια η εξουσία εδώ προφανώς είναι πάντα στα χέρια του εργοδότη με αυτές τις συμβάσεις μηδενικής εργασίας, αλλά φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με αυτές τις μηδενικές ώρες. Ε, μόνο εργοδότης καθορίζει πότε και για πόσο, μπορούν μόνο να δεχτούν τη σύμβαση και αυξάνεται ο κίνδυνο να μην ξανά υπάρχει εργασία και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και κίνδυνο να μην λαμβάνουν και κοινωνική ασφάλιση. Ε, πολλές φορές ε, οι υποστηριχτές ε, ε, που θέλουν να είναι ελεύθεροι εργασίες, ε, ε, να παρέμβουν στην αγορά εργασία, παρουσιάζουν αυτό ω μια ευέλικτη μορφή εργασία. Αυτέ όμω οι συμβάσει μηδενική εργασία χρησιμοποιούνται ευρέω και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχει καμία προστασία για τον εργαζόμενο και καμία ασφάλεια για την εργασία. Είναι η κατάχρηση λοιπόν τη εργασία των ανθρώπων αυτών και ορισμένε φορέ είναι πάντα στα χέρια του. Το 33% του προσωπικού στι συμβάσει μηδενικών ορών απασχολούνται για τουλάχιστον 6 μήνε και το 65% για 2 και παραπάνω χρόνια. Αυτέ οι συμβάσει μηδενικών ορών φαίνεται ε, ως ένας τρόπος να αποφύγουν τι ευθύνε των εργοδοτών παρά για να υπάρχει πραγματική ανάγκη για ευελιξία. Μόνο το 42% αυτών που έχουν συμβάσει μηδενική εργασία ε, λένε ότι έχουν δυνατότητα επιλογή. Ε, το 38% θα ήθελε να εργάζεται περισσότερο από ό,τι εργάζεται και ένα 14% λέει ότι αφού δεν έχει επαρκεί ε, ώρε για να εργαστεί ακόμα και το κατάλληλο βιωτικό επίπεδο, επίπεδο, δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο, το ενίκιο, ε, τους λογαριασμούς, ε, τρόφιμα κλπ. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη αύξηση στη χρήση των ε, τραπεζών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επιπλέον για αυτούς που αναζητούν θέση εργασίας ε, και ένα επιπλέον κίνητρο για τους εργοδότες είναι να προσφέρουν αυτές τις μηδενικές θέσεις εργασίας, διότι αν δεν λάβουν ε, αυτά τα, στις συμβάσεις δεν αποδεχτούν, θεωρείται κάποιος ότι δεν δέχεται μια θέση εργασίας και αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας διακόπτεται το επίδομα ανεργίας. Ε, υπάρχει λοιπόν πολύ μικρή δυνατότητα επιλογής σε, σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να δούμε καταρχάς τι ορολογία χρησιμοποιείται για να περιγραφούν αυτές οι συμβάσει μηδενικών ορού. Ορισμένες φορές ε, ε, εσκεμένα έχουν ε, προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το γεγονός είναι ότι αυτές οι συμβάσεις συνήθως πάντα προσφέρονται ε, με ε, μια, επί μια βάση ότι αν θέλεις, αν δεν θέλεις, μπορείς κάλλιστα να αποχωρήσεις και φυσικά υπάρχει και μια θεμελιώδης παρανόηση και διαφορετική παρουσίαση της δυναμικής σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργοζομένου. Ε, προτείνει το τι είναι ίση και ο εργοδότης ε, μπορεί να επιλέξει πώς θα απασχολήσει κάποιον. Πρόκειται για ένα πραγματικό μύθο για τους εργαζομένους. Ε, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι όταν συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις. Και επίσης όσον αφορά τη Σύμβαση Απασχόλησης ε, ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο όρο που χρησιμοποιείται και κάνει διάκριση μεταξύ των αυτοαποσχολουμένων και των ανθρώπων που εργάζονται με αυτές τις συμβάσεις. Πολλές φορές ε, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα πράγματα. Τώρα, η αξία του καθεστώτος του εργαζομένου δίνεται μια ψευδής επίφαση ότι ε, υπάρχει πραγματικά απασχόληση και πραγματικά ε, μπορεί έτσι κάποιος να λάβει δάνειο και να γνωρίζει ότι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ε, και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε ένα σύστημα επιδομάτων. Υπάρχουν όμως... Ε, εκτίματα, τους στερούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα που σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, έχουν το ίδιο καθεστώς υποτίθεται με τον αυτοαπασχολήμενο, αλλά αυτό δεν καλύπτει ούτε την επιθυμία του ανθρώπου, ούτε την πραγματικότητα. Στη... Ορισμένοι επιλέγουν απλώς να είναι αυτοαπασχολούμενοι, όπως ένας φυλακισμένος επιλέγει να παραμείνει στη φυλακή. Το γεγονό ότι δεν έχουν άλλε δυνατότητε επιλογή. Αν δείτε, για παράδειγμα, του αυτοαπασχολούμενου. Σκεφτείτε το Ίμπερ και το Deliveroo ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τι συμβαίνει με τι επιχειρήσει αυτέ. Ε, Ορισμένε φορέ ε, ο εργοδότης ε, μεταβιβάζει κάποιο από τον κίνδυνο της ε, διαχείρισης της επιχείρησης στον εργαζόμενο. Και ε, βάσει και του Ιδρύματος Resolution, ο μέσος μισθός είναι 12.000 λίρες το χρόνο. Και υπάρχει μια έκθεση το 2012 που λέει ότι το 40% των αυτοαποσχολημένων είναι ή στο ελάχιστο κατώτατο μισθό ή κάτω από αυτόν. Και πραγματικά είναι ελάχιστα τα κέρδη τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το γεγονό ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για τον εργαζόμενο είναι θεμελιώδες ε, ε, ζήτημα και ε, υπάρχει εδώ πέρα μια διατάραξη της ισορροπίας. Ε, οι εργοζόμενοι νιώθουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην δεσμεύονται τόσο με την επιχείρηση και να μην κάνουν την επιπλέον προσπάθεια. Ε, στο δικό μου το σωματείο, αν ένα εργαζόμενος δεν είναι διατεθειμένος να εργαστεί ως άτομο, γιατί να περιμένει ο εργοδότης ότι θα ε, δεσμευτεί με τον εργοδότη αν δεν του προσφέρει τα κατάλληλα πράγματα. Και ορισμένες φορές υπάρχουν και αμοιβέ υποχρεώσεις. Τώρα, ρήτρε αποκλειστικότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνηση έκανε μια διαβούλευση το 2013 και σε αποτέλεσμα αυτή διαπίστωσαν ότι το 9% των ατόμων που έχουν συμβάσει μηδενικών ωρών ουσιαστικά ε, βρίσκονται παγιδευμένοι σε ε, αποκλειστικέ συμβάσει εργασία ε, και ένα 15% μπορούσε να αναζητήσει σε κάποιε περιπτώσει μόνο θέσει εργασία. Και έχουμε και ένα 24% με κάποια μορφή αποκλειστικότητα ή κάποιο περιορισμό και ένα 39% μόνο δεν έχει επικλειστικότητα. Αυτές οι ρήτρε αποκλειστικότητας ουσιαστικά επιτρέπουν στους εργοδότες να έχουν και, το σκυλο... και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Ε, και υπάρχουν και κάποιες αναφορές στο Brexit ε, και δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα πράγματα και στρεβλώνουν και την πολιτική πραγματικότητα. Μπορεί να μην υπάρχει ανταγωνιστικότητα, δεν υπάρχουν δυνατότητα γνώσεων ε, και δεν μπορεί να καταβληθεί αυτό, διότι το κόστος επιβαρύνει ουσιαστικά τον, εργαζόμενο κάθε φορά. Οι ρήτρες αυτές αποκλειστικότητας θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα για πιο παραδοσιακές μορφές απασχόλησης και εκπαίδευσης ε, και επιμόρφωσης επιπλέον. Αυτές οι ρήτρες ε, αποκλειστικότητας ε, παρατηρείται ότι δεν δίνουν τελικά ωφέλη και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι χαμηλής απασχόλησης και κάνουν ε, θέσεις ε, χαμηλών ε, δεξιοτήτων, επομένως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζητήσουν και περαιτέρω επιμόρφωση. Το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει να υπάρχουν ε, διαιτησίες για την επίλυση διαφθοράς. Πιστεύω, κατά την άποψή μου γίνεται αυτό, διότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι έτσι θα φανεί δίκαιο. Δεν είναι πραγματική αυτή η δυνατότητα να προσφύγει κάποιος σε διαιτητικό δικαστήριο ο κώδικας διοντολογίας. Το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ε, απαντήσει ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας ε, για να υπάρχουν κάποιες ε, εξασφαλίσεις για αυτές τις συμβάσεις μηδενικής εργασίας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι κάθε ε, ε, σύμβαση εργασίας, θα πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες. Ε, υπαγορεύεται όμως η όρη από τους εργοδότες και οποιαδήποτε αθέμητη πρακτική θα μπορούσε έτσι όπως είναι γραμμένη και διατυπωμένη να φαίνεται σαν δίκαιη. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νομοθετημένες ε, ε, πρακτικές και δεν υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος να υποχρεώνει τον εργοδότη να συμμορφωθεί, ε, στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα για συνδοσία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανισμός εφαρμογής δεν δίνει καμία δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο, μπορεί απλώς να αρνηθεί και όταν βρίσκονται σε τέτοιες επονίδιστες συνθήκες δεν έχουν και άλλη λύση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία άλλη λύση παρά να δεχτούν ακόμα και αυτές τις ρήτρε της αποκλειστικότητες. Ε, υπάρχει χρήση και κατάχρηση λοιπόν αυτών των συμβάσεων μηδενικών ορών εργασία. Και πιστεύετε ότι ε, δεν είναι ανοησία, αλλά αυτό γίνεται μόνο από αυτού οι οποίοι θέλουν να νομιμοποιήσουν αυτές τις πρακτικές. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τα εξής ε, από εδώ και πέρα. Όλε οι συμβάσει μηδενικέ εργασίες θα πρέπει να θεωρούνται συμβάσει απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι θα ασκείται ε, το εργατικό δίκαιο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 23 του εργατικού δικαίου από το 1999 που καθορίζει συγκεκριμένα ο καθεστώ απασχόληση για όσου έχουν σύμβαση εργασία. Έτσι θα αρθούν και οι αβεβαιότητε και θα υπάρχουν και ε, ε, έλλειψη κινήτρων για κάποιου αδίστακτους εργοδότες και επίσης θα μπορούσε να υπάρχει κάποια αρρύθμιση ώστε μετά από κάποιο διάστημα εργασίας με σύμβαση μηδενικών ωρών να μπορεί κάποιος να το μετατρέψει σε μόνιμη σύμβαση εργασίας. Αυτό προβλέπεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο για αυτούς οι οποίους έχουν σύμβαση ορισμένου ε, χρόνου για ένα συνεχές διάστημα τεσσάρων ετών, χωρίς να προτείνουμε οπωσδήποτε ότι θα πρέπει να είναι τέσσερα χρόνια. Ο εργαζόμενος ε, με μηδενικές ώρες εργασίας έτσι δεν θα βρίσκεται σε θέση ε, να κάνει κατάσταση κατάχρηση της σύμβασής του ο εργοδότης του. Ε, υπάρχει και μια οδηγία η οποία βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων και καλύπτει ε, τα θέματα αυτά και λέει ότι το μέτρο του δυνατόν οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα των εργαζομένων να μετατρέπουν τις συμβάσεις ε, ή να αυξάνουν το χρόνο εργασίας όταν προκύπτει τέτοια ευκαιρία. Επειδή οι μηδενικές ε, ώρες εργασίας είναι μορφή μερικής απασχόλησης, μπορεί να καλύπτονται και από αυτή τη διάταξη. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που καθορίζουν το χρόνο εργασίας εργασία, όχι μόνο το χρόνο κατά τον οποίο εργάζεται, αλλά και το χρόνο που είναι διαθέσιμος στο ή κοντά στο χώρο εργασίας. Και με αυτό θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην ε, Κέρστιν Χάουαλτ. Για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τους ε, εργαζόμενους στην ε, γεωργία, τον τουρισμό και την, τα τρόφιμα. Ε, να σας μιλήσω για τα fast food, τα ταχυφαγεία. 700.000 εργαζόμενοι, 225.000 μόνο στο McDonald's. 1,9 εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος εργαζόμενος σε όλο τον κόσμο. Τα χαρακτηριστικά, όπως γνωρίζετε, είναι ότι είναι, οι εργαζόμενοι είναι νέοι, πάνω από το 50% είναι κάτω των 25 ετών, στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από το 42% κάτω των 21 ετών. Πολλοί φοιτητέ, γυναίκες, μετανάστευς, ε, πολλά άτυπα, πολλές άτυπες συμβάσεις εργασίας, ε, ε, προσωρινή εργασία, περιορισμένου χρόνου κλπ. 60-70% στον Βασίλειο είναι ε, περιορισμένου χρόνου και πάρα πολλοί από αυτούς ε, σε, με συμβάσεις ε, μηδενικού χρόνου. Πολύ λίγοι μένουν παραπάνω από ένα χρόνο. Πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικέ συμβάσει, ένα ε, τομέα πολύ δύσκολο να συνδικαλιστεί, πολύ χαμηλή εκπροσώπηση, μικρή συμμετοχή σε συνδικάτα. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη εναλλαγή στο εργατικό δυναμικό και όπως σας είπα και το 80% ε, αυτών των ε, καταστημάτων είναι καταστήματα δικαιώχρησης, franchise. Οπότε η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πάρα πολύ ακριβή στοιχεία. Αυτά είναι που σας είπα τα βασικά στοιχεία που έχουμε για το τομέα του fast food. Για τις τρεις αναφορές ο Ιαν ε, περιέγραψε πολύ καλά την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να σας πω ότι γίνεται στο Βέλγιο. Έχουμε τα ε, ελαστικά συμβόλαια, flexi jobs. Ε, το νομοσχέδιο το οποίο θετήθηκε στο τέλος 15 για αυτά ακριβώς τα συμβόλαια οδήγησε τα συνδικάτα στο να προσφύγουν στο συνταγματικό δικαστήριο προκειμένου να καταργηθεί το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε το τέλος Σεπτεμβρίου να μην το καταργήσει το νόμο. Η χρήση αυτών των συμβάσεων ε, ξεκίνησε στον τομέα της εστίασης και του ξενοδοχειακού τουρισμού. Ε, ο αριθμός αυξήθηκε πάρα πολύ σε ένα χρόνο. 500% αύξηση από το 2015 στο 2016 στη χρήση τέτοιων συμβάσεων. από 2.000 σε 20.000 το χρόνο. Ε, αυτοί οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται για τις διακοπές τους, δεν χαίρουν συλλογικών συμβάσεων, έχουν χαμηλότερους μισθούς κλπ. Και το κακό είναι ότι αυτά, αυτές οι συμβάσεις θα διευρυνθούν, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στο Βέλγιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ερευνητές, την Αριστεία και τον Γιάννη για την πολύ βαθιά, σε βάθος ανάλυση των αναφορών που ε, αφορούν τα ταχυφαγεία. Συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας και τις προτάσεις σας. Οι άτυπες μορφές εργασίας ε, αποτελούν μετακίνηση του κινδύνου από τον εργοδότη στον εργαζόμενο και αυτά συνοδεύονται επίσης και με άλλα θέματα ε, όπως η φόρο αποφυγή. Το βλέπουμε και σε διασυνοριακό επίπεδο σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά βλέπετε ότι αυτό ισχύει και για μικρότερες επιχειρήσεις. Συμφωνώ επίσης με τα συμπεράσματά σα για το, την ανάγκη να ε, γεφυρώσουμε τα κενά, να καλύψουμε τα κενά που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Κοινωνική και Εργασιακή. Χρειαζόμαστε δικαιώματα για όλους, ίση μεταχείριση σε όλους ανεξαρτήτως ε, του καθεστώτος υπό το οποίο εργάζονται και ανεξαρτήτως της σύμβασης εργασία τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους αυτοπασχολούμενους, ε, αλλά και τις, τους εργαζόμενους στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Νομίζω ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν σύμβαση ε, και κοινωνική κάλυψη από τουλάχιστον την πρώτη μέρα της εργασίας τους. Αυτό θα ήταν ένα καλό εργαλείο, ένα καλό πρώτο βήμα. Για να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις ατυπ, ατυπές ε, ή επισφαλείς ε, μορφές εργασίας. Και να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια στους εργαζόμενους. γιατί όχι και μια συμφωνία πλαίσιο, μια οδηγία πλαίσιο για αυτό το θέμα. Επίσης, ε, ε, ελπίζουμε ότι οι αναφορές και το έργο της Επιτροπής Αναφορών θα βοηθήσουν στο να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε στόχο μια κοινωνική Ευρώπη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που εξοικονομήσατε και κάποιο χρόνο. Ε, αυτό πάντα το επικροτεί ένας πρόεδρος. Ε, ε απευθύνομαι αμέσως στον ε, διπλανό σας, τον κύριο Ντεμικέλε. Δέκα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας. Ehm, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παρέμβασή μου Ε, την οποία συνέλεξα από την ε, μακρά ε, έκθεση που άφησα στη διάθεση της Επιτροπής Αναφορών κατόπιν της αναφοράς, εξέτασα την Ευρωπαϊκή Νομολογία για τις δύο ρήτρε της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 70 του 1999 για την εργασία ορισμένου χρόνου. Εξετάζοντας όλη την ομολογία και ε, εν ώψη και συμμετοχής ε, σε κάποιες ε, υποθέσεις στο δικαστήριο και πιο συγκεκριμένα σε ιταλικές υποθέσεις, προκύπτει αμέσως ένα ανησυχητικό πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο εκφράζεται μέσω της ποιότητας και του αριθμού των αναφορών που είναι ακόμα ανοιχτέ ε, εδώ στην Επιτροπή σας. Η τεράστια πλειοψηφία των αποφάσεων και των ε, ε, επιταγών του ε, δικαστηρίου για τη ρήτρα 4 για την μη διάκριση μεταξύ ε, των συμβάσεων ε, ορισμένου και αορίστου χρόνου και για τον άρθρο 5, δηλαδή αυτό το οποίο προβλέπει τα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για παρεμβάσεις και για κυρώσεις πιθανών σε περίπτωση κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου αφορούν τις δημόσιες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, Εάν ε, δεν είχε υπάρξει η πρώτη καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η καταδίκη Μάγκολτ ε, του ε, του Οκτωβρίου του 2005, ε, μία απόφαση η οποία δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα για μία ανύπαρκτη υπόθεση. Πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο δημιούργησε και μία σειρά από πολύ δυσάρεστες συνέπειες και για το δικαστήριο και για κάποιες χώρες και τις αντιδράσεις προτάσεις που είχαν, πιο συγκεκριμένα η Γερμανία, για τη λύση την οποία επέκρινε το ίδιο το δικαστήριο και επέλυσε στη συνέχεια με μια μελλοντική απόφαση Αντενέρ, χωρίς να υπήρχε λοιπόν αυτή η απόφαση Μάγκολτ. Και την άλλη απόφαση ε, Deutsche Lufthansa σε σχέση ε, ε, με τις ιδιωτικές θέσεις εργασίας, αυτή τη στιγμή θα υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο μόνο για αποφάσεις του δικαστηρίου που αφορούν απλώς και μόνο ε, επικρίσεις για τη χρήση ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τις δημόσιες αρχές. Ποιών κρατών μελών. Εγώ εδώ έχω σχεδόν 10 χώρες. Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Ισπανία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ρουμανία. Όλες αυτές οι χώρες ε, ε, είχαν σχετικές προσφυγές από ε, προδικαστικά ερωτήματα τα οποία έθισαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφορούσαν δημόσιες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε το εξή. Εάν ε, η μεγάλη πλειοψηφία των αναφορών που συζητούνται από εσά εδώ σήμερα αφορούν ε, τι επισφαλεί θέσει εργασία ε, του δημοσίου τομέα, πέραν των συμβάσεων με μηδενικέ ώρε εργασία που έχουν επινοήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά που έχει και τις καταβολές του στην Ιταλία. Στην Ιταλία υπάρχει αυτή η εποχική εργασία, η οποία βασίζεται στην ίδια λογική. Κάτι λοιπόν δεν έχει πάει καλά στον έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας 9970. Ε, Διότι η χώρα δεν μπορεί το κράτος μάλλον δεν μπορεί να υπερασπιστεί ε, αυτόν ως δημόσια διοίκηση αν δεν εφαρμόζει ε, την οδηγία 9970. Υπάρχει μια οριζόντια και κάθεται όμως εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Αν όλες οι χώρες είχαν τη δυνατότητα ως εργοδότες να αποφύγουν να εφαρμόσουν την οδηγία, τότε προφανώς ε, η οδηγία δεν θα είχε κανένα νόημα. Και ε, πράγματι το πρόβλημα από όλε αυτές τις αποφάσεις του δικαστηριού και από όλε αυτές τις ε, ε, καταδίκες είναι το εξής, ότι η οδηγία 9970 δεν εφαρμόστηκε όσον αφορά περιπτώσεις δημόσιας διοίκησης. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα όργανο το οποίο αποκαλείται Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στόχο έχει να μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή των συνθήκων. Αντί λοιπόν απλώς να αναρωτιόμαστε εάν πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία 9970, όπως ορισμένες φορές αναρωτιόμαστε και εμείς στην Ιταλία όταν πρόκειται για τροποποίηση του συντάγματός μας, ε, και μετά τίθεται η περαιτέρω ερώτηση. Μήπως ε, δεν έγινε εφαρμογή στο συγκεκριμένο τμήμα του Ιταλικού Συντάγματος. Μήπως λοιπόν δεν έχει γίνει εφαρμογή της 9970. Η οδηγία 9970 δεν εφαρμόστηκε ε, και αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων και η ποιότητα μίας εκ των αναφορών που ε, παρουσιάστηκε εδώ σε εσάς. 108 συμβασιούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε φορά που πρόκειται για εφαρμογή του άρθρου 5, δηλαδή τα προληπτικά μέτρα, τα ε, ε, μέτρα κατάχρησης ε, κατά των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαφανίζεται. Στις αποφάσεις στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια λαμβάνει απόφαση αμφίσιμη στη συνέχεια. Δηλαδή, δεν θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεν έχουν συμμορφωθεί στην οδηγία, ενώ ταυτόχρονα καθορίζουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια εφαρμογής, τα οποία δημιουργούν επισφάλεια. Εμείς ήμασταν ε, μάρτυρας μόνο μίας ε, προσφυγής ε, για μη συμμόρφωση της οδηγίας κατά του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η συγκεκριμένη προσφυγή, η οποία οδηγήσε στην απόφαση της 20ης της Φεβρουαρίου του 2015 κατά του Δουκάτου του Λουξεμβούργου, γιατί δεν συμμορφώθηκε προς την οδηγία 9970 για μια πάρα πολύ περιορισμένη ε, μερίδα εργαζομένων, των επισφαλών εργαζομένων στο χώρο του θεάματος και μόνο και τότε μόνο υπήρχε παρέμβαση για μη μόρφωση προς την οδηγία και αυτό είναι καρπός ε, τα όσα έγιναν στις 7 Μαΐου του 2014. ήμουν παρόν και επομένω μπορώ να σας πω απευθείας τι συνέβη όταν διαμαρτυρηθήκαμε ως Ιταλοί νομικοί ότι ενώ συζητούσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους αντικειμενικούς λόγους ως προληπτικό μέτρο κατά της ε, διαδοχής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δηλαδή υποστηρίζαμε τη θέση που υποστήριζε και το δικό μας ακυρωτικό δικαστήριο ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν ο κανόνας και οι συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν η εξαίρεση, τότε όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση, ο Εθνικός Δικαστής συγγνώμη, ο κοινοτικό δικαστή διορθώνει ο μιλητή, όταν ε, ε, αντιλήφθηκε ότι από εκείνο το προδικαστικό ερώτημα ο εθνικό νομοθέτη είχε δημιουργήσει μια νομοθεσία που απαγόρευε οποιαδήποτε μορφή προστασία, εμεί ε, διαμαρτυρηθήκαμε ε, επισήμω. Παρενέβη ο δικαστή Τότερ που συμμετείχε τότε στο τρίτο τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση κατά της Ιταλίας για το Jobs Act ε, ξεκίνησε τη διαδικασία για τη μη συμμόρφωση προς την οδηγία κατά το δικά του Λουξεμβούργου. Εδώ στην Επιτροπή αναφερών πολλές φορές όσον αφορά για τις ε, αναφορές ε, για τα σχολεία. Υπάρχει και μια αναφορά ε, για έναν υπάλληλο της υπηρεσίας εισόδων που ε, αρχιοθετήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών απλώς για τον μόνο λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και σας παρουσίασε μία κατάσταση που δεν θεωρείται ότι είναι κρίσιμη για σχέση για τη συγκεκριμένη αυτή. Έδωσε ψευδείς ε, πληροφορίες στην Επιτροπή Αναφορών για μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, την απόφαση Μάρκο Τσαμοάνο, η οποία έλεγε ε, ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο σας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η κατάσταση είχε πάρα πολύ σοβαρέ συνέπειε όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, για παράδειγμα των υπαλλήλων ε, σε αυτή την υπηρεσία. Διότι υπήρχε απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου του 2015 που έλεγε ότι δεν εφαρμόζονταν επαρκώ η οδηγία. Ήταν πλημελή η εφαρμογή τη. Και αλλάζει η κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι η Επιτροπή Αναφερών ε, την έκλεισε τη διαδικασία επιπαραβάση. Στην ουσία ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία είπε ότι πρέπει να κλείσετε την υπόθεση γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και άλλαξε την ομολογία σε σχέση ε, με αυτούς τους υπαλλήλου, και έτσι η οδηγία δεν εφαρμόζεται. Και εμείς στην Ιταλία φτάσαμε στο εξή σημείο ο δικαστής και υπάρχουν πάρα πολλές ε, αναφορές οι οποίες ε, παρουσιάστηκαν εδώ. Οι δικαστές λοιπόν δεν θε, λαμβάνονται και δεν θεωρούνται καν ε, εργαζόμενοι γιατί δεν εφαρμόζεται η οδηγία 9970. το άρθρο 4 και το άρθρο 5 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξετάζει για να προστατεύσει τα προσωπικό της συμφέροντα, δηλαδή τη, το, τους συμβασιούχους που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ότι δεν ισχύουν. Και φτάνω στα συμπεράσματά μου. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, σε μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει μια εξωσυμβατική πάρα πολύ σοβαρή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν φρόντισε για την σωστή εφαρμογή της οδηγίας 9970, ε, ε, ε, σημαίνει ότι η Επιτροπή Αναφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρέμβουν. δάλους θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ βαριά ε, διαδικασία με πάρα πολλούς επισφαλείς ε, εργαζομένους στο δημόσιο τομέα και θα υπάρχουν ε, και πολύ σοβαρές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν καλύπτει τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται για αυτήν από την Ευρωπαϊκή από την συνθήκες. Very... Σας ευχαριστώ πολύ πολύ ισχυρά και σαφή τα μηνύματα της παρεμβασής σας. Δίνω τώρα το λόγο στους δύο τελευταίους ομιλητές που εκπροσωπούν αναφέροντες. Για πέντε λεπτά ο κύριος Γκαλεάνο και μετά ο κύριος Άσπουκ. Παρακαλώ. Ε, οι προηγούμενοι ομιλητές παρουσίασαν κάποια προβλήματα ε, στον τομέα της επισφαλούς εργασίας, αλλά από όσα είπε και ο δικηγόρος Δεμικέλε που μίλησε πριν από μένα, υπάρχουν και ε, στοιχεία στην έκθεση Eurofound, κυρίως ε, για τον ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Δεμικέλε, το σημαντικό αφορά τις θέσεις του δημοσίου τομέα, ιδίως στην Ιταλία. Ένα τομέα στον οποίο στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα από την κρίση του 2008, διότι οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στους Ευρωπαίους πολίτες ε, ε, ε μειώθηκαν ε, σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Όσον αφορά τις αναφορές που εκπροσωπώ εγώ σήμερα, είχαμε την έκθεση 2007-2008 ε, το επισφαλές προσωπικό της Ιταλίας ουσιαστικά είναι περίπου 290.000 άνθρωποι. Στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας ε, ε, είναι πάνω από 30.000 άνθρωποι. Ε, πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν εκπροσωπούν καταλήλω. Τα στοιχεία είναι πολύ μεγαλύτερα. Κυρία Πρόεδρε, αυτή τη θέση δεν τη λέω εγώ υποκειμενικά. στο πίνακα, στο σημείο 5.5 στην έκθεση, έχουμε 10.392 επιφαλείς εργαζόμενους ε, σε περιφέρειες οι οποίες είναι ειδικού ενδιαφέροντος στην Ιταλία. Στη Σικελία, που είναι μία από τις πέντε περιοχές που θεωρούνται ειδικού ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι είναι η πιο μεγάλη, όπως φαίνεται από την έκθεση του 2015 στον ε, επιθεωρητή εργασίας ε, που ασχολείται με τα θέματα αυτά, οι επιφαλείς εργασίας είναι 16.798, στις οποίες προτίθενται 5.410 εργαζόμενα, οι οποίοι υποπληρώνονται και δεν έχουν κατάλληλη κοινωνική ασφάλιση. Επομένως, συνολικά, μόνο στη Σικελία από τις 5 αυτόνομες περιοχές έχουμε 22.168 επισφαλείς εργαζομένους που είναι πάνω από το διπλάσιο αυτών που αναφέρονται στην έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Ιταλίας. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους τομείς θεωρούμε και αυτό που είναι ουσιαστικό είναι ότι στον τομέα της υγείας ότι μεγαλύτερος αριθμός ε, των ανθρώπων που εργάζονται στις επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι νοσοκόμοι. Ε, αλλά υπάρχουν και οι ιατροί που εργάζονται και που πολύ συχνά υποδεικνύονται ως ελεύθεροι εργαζόμενοι ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται κανονικά ως μισθωτοί. Ε, με τέτοια λοιπόν στοιχεία δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι οι επισφαλείς εργαζόμενοι είναι κατανομημένοι σε όλη την δημόσια διοίκηση της Ιταλίας αλλά και σε όλη την Ιταλία και από τη Σικιαλία, από τους επισφαλείς εργαζομένους της Ιταλίας ακόμα και στη Βάλεντα Όστα ε, που ε, αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2015 που αφορά τους επισφαλείς εργαζομένους της Βάλεντα Όστα που βρίσκεται στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία η περίοδος επισφαλούς εργασίας ε, υπερβαίνει τους 36 μήνες που είναι το εσωτερικό όριο που έχει θέσει το Ιταλικό κράτος ε, για τις ε, συμβάσεις επισφαλούς εργασίας, ορισμένου χρόνου, συγγνώμη, και ορισμένες φορές μπορεί να φτάνει τα 20 και 25 χρόνια. Και εδώ η κρίση του 2008 δεν έχει καμία σχέση φυσικά με το πρόβλημα το μέγιστο όριο το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία είναι 36 μήνες. Αλλά ε, το γεγονός ότι ξεπερνιέται αυτό το όριο δεν σημαίνει ότι σταθεροποιείται ο, ο επισφαλής εργαζόμενος στην Ιταλία γιατί υπάρχει το θέμα του διαγωνισμού. Και μάλιστα σε μια κατάσταση στην οποία οι διαγωνισμοί δεν γίνονται ποτέ ε, στο σχολείο όπως ε, διαπιστώνεται από την απόφαση Μάσκολο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Νοεμβρίου του 2014 στον σχολικό τομέα από το 1999 μέχρι το 2012 δεν έγινε κανένας διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και για την αυτόνομη περιοχή της Σικελία, όπου ε, εδώ και 30 χρόνια δεν γίνονται διαγωνισμοί του δημοσίου. Ε, ενώπιον λοιπόν αυτής της κατάστασης διαπιστώνεται ότι ε, η μονιμοποίηση στους ε, καταλόγους μετά ε, από τις 30.000 ε, ανθρώπους που ε, προσελήφθησαν το 2007-2009 με το λεγόμενο νόμο πρώτη του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγιναν μετά από την απόφαση του δικαστηρίου Μορόζο Σαρντίνο και μετά από εκεί και πέρα μειώθηκαν σε κάποιες χιλιάδες για τα επόμενα χρόνια. Από εκεί διαπιστώνουμε πολύ εύκολα ότι στην πραγματικότητα ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αλλά και οι άλλες ευέλικτες συμβάσεις χρησιμοποιούνται για να καλύψουν θέσει ε, στη δημόσια διοίκηση που θα έπρεπε να είναι μόνιμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κενέ. Και αυτό σε ένα τομέα τη δημόσια διοίκηση, όπου έλεγα ότι ε, επηρέασε πολύ λίγο η ε, κρίση, διότι απλώ. σταμάτησαν οι αυξήσεις του μισθούς για πέντε χρόνια. Ε, ενώ δεν μειώθηκαν θέσεις εργασίας. Ε, επομένως, διαπιστώνουμε ότι και σε οργανωτικό επίπεδο ε, και στο δικαστικό σώμα 5.000 τακτικοί δικαστές οι οποίοι βρίσκονται και στους, με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει και μια εμβληματική υπόθεση των πρώην εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για πάνω από 20 χρόνια για να καλύπτουν νέες θέσεις μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου ακριβώ γιατί δεν είχε διεξαχθεί διαγωνισμό και εργάζονταν σε θέσει που θεωρούνται κενέ. Ε, και φυσικά ε, υπήρχε και τεράστιο πρόβλημα φοροδιαφυγή. Ε, ακριβώς λόγω αυτού του φαινομένου. Σε μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ε, υπάρχει νομοθεσία ε, του Μαΐου του 2017 της Ιταλίας, αλλά η νομοθεσία αυτή είναι πλήρως ανεπαρκής. Αφορά μόνο το 50% των διαθέσεων θέσεων εργασίας, αφορά κάποιους που έχουν πάνω από 15 χρόνια επισφαλούς θέσεων εργασίας και αφορά μόνο συγκεκριμένου χρήστε και δεν υπάρχει υποχρέωση για συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων. Καλύπτει λοιπόν εν μέρη και μάλιστα σε πολύ μικρό βαθμό το πρόβλημα των επισφαλών εργαζομένων στην Ιταλία. Ολοκληρώνω σιγά σιγά. Εδώ θα πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η επισφαλή κατάσταση έχει πολύ συμβαβαρέ συνέπειε για χιλιάδε ανθρώπου, όχι μόνο για ψυχολογικού λόγου, αλλά το γεγονό ότι βρίσκονται σε έλλειψη ασφάλεια αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν για παράδειγμα ένα δάνειο για αγορά πρώτη κατοικία ε, και δεν μπορούν να ζήσουν έτσι αυτόνομα και να δημιουργήσουν οικογένεια. Για να μην δεν μιλήσω για τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά. Πρόκειται για κατάσταση τις οποίε ο Ευρωπαίος νομοθέτη είχε εγκρίνει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999-70. Ε, ζητούμε λοιπόν, καλώντας ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ελέγξει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί να τροποποιήσει την οδηγία, να φροντίσει για την εφαρμογή της. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που ε, σας πιέζω ως προς το χρόνο. Δεν ε, θα, θα προτιμούσα να μην το κάνω, αλλά ο, ε, μας περιορίζει ο χρόνος. Προχωρώ κατευθείαν στον Μάικλ Άσπρουκ που εκπροσωπεί τους συμβασιούχους υπαλλήλους. Θα προσπεράσω όσο γίνεται περισσότερες από τις διαφάνειες μου για να γλιτώσουμε χρόνο. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τις πάρετε από την ΠΕΤΗ, ε, από μένα προσωπικά, από την ιστοσελίδα ΣΥΝΤΗ και μάλιστα ε, μέσα σε μια ώρα μπορείτε να την πάρετε πλάστο Λουξεμβούργ 8 και να μου αγαράσετε και ένα ποτό, να με κεράσετε ένα ποτό. Ζητώ συγγνώμη, έχει κολλήσει το μηχάνημα. Α, σας παρακαλώ μην το αφαιρέσετε αυτό από το χρόνο μου. Έχει κολλήσει το σύστημα. Ah, that's very kind. Ah. Α, ωραία. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όχι, δεν λειτουργεί. Να βλέπετε, αυτά είναι τα αποτελέσματα της λιτότητας. Όλα καταραίουν. Brief. What are we going to do? What are we going to do? Τι θα κάνουμε? Can I get there? Μπορώ να έρθω να καθίσω εκεί. oh, sorry. Uh, Madam Chair. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, εκπρόσωποι των μίδια, ε, πολίτες ε, και ε, επίσης αγαπητοί φίλοι σε επισφαλής εργασίας. Το να απολύει κανείς ε, κάποιον αυτομάτως ε, μετά από έξι χρόνια με τη μεγάλη πείρα που έχουν αποκτήσει ε, στο μεταξύ αποτελεί μεγάλη σπατάλη. Ελάχιστες εταιρείες θα το κάνανε αυτό. Ε, κάποιος που εργαζόταν μια χαρά επί έξι χρόνια ξαφνικά δεν μας κάνει πια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγωνίστηκε σκληρά για να αρνηθεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, από τους ε, ε, υπαλλήλους της. Μάλιστα, το... υπήρχε η αντιδικία με τον κύριο Στράκ. Ο κύριος Στράκ όμως τελικά κέρδισε την διαμάχη η οδηγία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ε, διέπουν, διέπει τις, ε, αυτές τις εργασιακές ε, σχέσεις. και γενικά πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές αυτής της οδηγίας. Έχουμε την αρχή των μη διακρίσεων. Όσον αφορά τη δεοντολογία, τι να σας πω, είναι αβυσαλαίο το πρόβλημα αν σκεφτεί κανείς ε, τι κάνει η Κομισιόν στους υπαλλήλους της ε, ξεχάστε σπίτι. Στο Λουξεμβούργο δεν πρόκειται να αποκτήσετε εάν ε, είσαστε συμβασιούχος. Μάλιστα θα είναι πρόβλημα ακόμα και η ενοικίαση μικρού διαμερίσματος, ε, διότι ε, οι ενοικιαστές ε, δεν θέλουν ανθρώπους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι θα εισπράξουν το νίκη. Φανταστείτε λοιπόν τι κάνει αυτό στα παιδιά σας. Ένα πολύ σημαντικό αίτημα είναι οι εσωτερικοί διαγωνισμοί να ανοίξουν και για τους συμβασιούχους υπαλλήλους. Ε, κάποιοι άνοιξαν το 2016 και κάποιοι συμβασιούχοι υπάλληλοι ε, έχουν αποκτήσει τώρα μόνιμες ε, θέσεις απασχόλησης, αλλά εμείς θέλουμε σύμφωνα με την οδηγία να ανοίξουν οι διαγωνισμοί αυτοί ε, απολύτως ε, για τους ε, συμβασιούχους, όπως είναι ανοιχτοί οι διαγωνισμοί και για τους μόνιμους υπαλλήλους. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το 25% των ανθρώπων αποκτούν μια θέση μέσω των εσωτερικών διαγωνισμών και μόνο το 1% με εξωτερικούς διαγωνισμούς. Και ε, ποια είναι η γενικότερη εικόνα. Η Ευρωβουλευτή Κέρτον Τάρλινγκ ε, αναφέρθηκε σε αυτό. Εξετάζουμε την πολιτική πτυχή του θέματος. Το θέμα των ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου υπονομεύει την Ένωση, υπονομεύει της Επιτροπής Προσεπικού και ένας από τους λόγους για την εξάπλωση του ακροδεξιού λαϊκισμού είναι κατά τη γνώμη μου ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται μη χάσουν και ε, γι' αυτό δεν μπορούν ε, να αγωνιστούν, ε, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο απλά να αποκλείσουν τους μετανάστες. Και κάτι ακόμα που θέλουμε είναι ίση πρόσβαση στην εσωτερική αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τους συμβασιούχους. Όλες οι θέσεις ε, θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμες ε, για τους συμβασιούχου. Τι ζητάμε, δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα, θέλουμε πιο πολύ σεβασμό, καλοσύνη και δικαιοσύνη. Σα ευχαριστώ και θα τα πούμε Πλάσου Λουξεμβούργκ, ε, ε, 8. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Άσπρουκ ε, νομίζω πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούω κάποιον να κλείνει ομιλία καλώντας ε, ε ανθρώπους να πιούν ένα ποτό. Απαντήσεις τώρα στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες ε, που τέθηκαν. Ε, έχουμε εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω πέντε λεπτά στον καθένα σας για να απαντήσετε. Εάν θέλετε να μοιράσετε διαφορετικά το χρόνο μεταξύ σας, μπορείτε να το κάνετε. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ποκόρνη από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση τμήματα αρχής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Αναφορών που διοργάνωσε αυτή τη σημαντική ακρόση όπως είπατε και στην αρχή, είναι πολύ επίκαιρη μάλιστα. Δύο μέρες περίπου, ελάχιστες μέρες, εν πάση περιπτώσει, μετά την απόφαση για το κοινωνικό πυλώνα του Γκάτεμπορκ. Ένας από τους βασικούς στόχους του κοινωνικού πυλώνα είναι να μειωθεί η επισφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώθει η πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να εστιάσω σε, στις δύο βασικές προσεγγίσεις ε, τις οποίες ακολουθούμε εμείς στο δικό μου κομμάτι της Κομισιόν για αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, είναι μέσω της εφαρμογής των ισχυουσών οδηγιών, για παράδειγμα την οδηγία για ε, τις ε, συμβάσεις ε, περιορισμένου χρόνου και δεύτερον η ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα. Υπάρχουν τρεις οδηγίες που έχουν σχέση με, την, ε, ε, με το πρόβλημα αυτό, η οδηγία περιορισμένου χρόνου, ε, η οδηγία μερικής απασχόλησης και η οδηγία προσωρινής απασχόλησης. Προσπαθούν να βελτιώσουν και οι τρεις οδηγίες αυτές την προστασία των εργαζομένων ταυτόχρονα προστατεύοντα την έννοια της ελαστικότητας που μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο στην δημιουργία θέσεων εργασία. Και οι τρεις ε, αυτές οδηγίες ε, έχουν ως ε, επίκεντρο την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει στο παρελθόν καταδικάσει τις διακρίσει ε, ανάμεσα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ή μόνιμης εργασίας και τις άλλες. Αυτό, αυτές οι διαφορές μπορούν να αφορούν και το μισθό και τα συνταξιδοτικά δικαιώματα, τις πολιτικές απολύσεων, ε, δυνατότητες προαγωγής, συμμετοχή σε αξιολόγηση ή σε κατάρτιση, καθώς επίσης και στο θέμα της αποζημίωσης που θα πληρωθεί σε περίπτωση απόλυσης. Ε, η δεύτερη διάταξη την οποία θα πρέπει να δούμε στην οδηγία των, του εργασίας περιορισμένου χρόνου είναι το να αποφευχθεί η ανανέωση, η επαόριστον ανανέωση αυτών των συμβάσεων αν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Αλλιώς θα πρέπει να υφίσταται ένα μέγιστος χρόνος ή μια μέγιστη, ένας μέγιστος αριθμός ανανεώσεων. Ε, θέλουμε αυτές οι οδηγίες να εφαρμόζονται όπως το πρόβλημα στο δικαστήριο και οι ίδιες οι οδηγίες, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής, ποιος καλύπτεται. Αυτό είναι ένα όλο και πιο προβληματικό ζήτημα. Ε, δεδομένου ότι υπάρχει μια ε, αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το ποιος είναι αυτοπασχολούμενος, ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος μισθωτός. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με την οδηγία ε, των συμβασιούχων, οι οποίοι δεν καθορίζονται με τρόπο πάρα πολύ ξεκάθαρο. Παρόλο που η οδηγία παραπέμπει εθνικές, στους εθνικούς ορισμούς και μάλιστα για τον πρώτο τελευταίο μιλητή να πω ότι το δικαστήριο σύντομα θα κρίνει την περίπτωση των ε, επίτιμων δικαστών στην Ιταλία και εκεί θα δούμε αν εμπίπτουν στην, στο πεδίο της οδηγίας ή όχι. Δεύτερον, ποιοι είναι συγκρινόμενοι εργαζόμενοι ε, για να αποφευθούν οι διακρίσεις. Μερικές φορές είναι δύσκολο με να ξέρουμε ποιους θα πρέπει να συγκρίνουμε. Μερικές φορές γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τύπους ε, συμβολέων, συμβάσεων περιορισμένης, ε, περιορισμένου χρόνου. Επίσης, ε, τι μπορεί να ε, επιτρέψει να έχουμε διαφορές σε, διαφορε, σε διαφορετικές, διαφορές ό,τι αφορά διαφορετικές συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ή ε, στην ίδια σύμβαση σε διαφορετικές ανανεώσεις. Πάντως, οι, περιορισ... συμβάσει περιορισμένου χρόνου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίζονται, να καλύπτονται ανάγκες μόνιμες. Τέλος, τι είδου ε, αποζημιώσεις ή ε, προσφυγές ε, έχουν οι εργαζόμενοι στα... στη διάθεσή τους σε περίπτωση που αδικηθούν. Προφανώς δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει δικαίωμα αυτόματης μετάβασης σε μόνιμη σύμβαση αλλά ε, υπάρχουν δυνατότητες προσφυγής. Και μάλιστα πολλές αναφορές, ιδιαίτερα από την Ισπανία και την Ιταλία, ε, έχουν κατατεθεί εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, συνεχίζουμε να εξετάζουμε το θέμα της, των ταχυφαγίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και το θέμα του Βελγίου Έχουμε έρθει σε επαφή με τα δύο αυτά κράτη-μέλη και όταν πάρουμε την απάντησή τους θα την αναλύσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Οι Ιταλικές ε, περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν εδώ ε, τις αναλύουμε αυτή τη στιγμή, αναλύουμε ένα νομοθετικό διάταγμα το οποίο θετήθηκε στην Ιταλία το καλοκαίρι και θα απαντήσουμε στην, για την ουσία της υπόθεσης στην Επιτροπή σας. Να δούμε αν θα πρέπει να ε, ξεκινήσουν διαδικασία επί παραβάση. Επίσης, ε, ό,τι αφορά το, την περίπτωση Σαντόρο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε ε, την, ε, το θέμα της, ε, κάποια ζητήματα σχετικά με την αποζημίωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερη προσέγγιση για τον κοινωνικό πυλώνα, ε, θα νομοθετήσουμε, αυτή τη στιγμή διαβουλευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους, μετά από αυτή τη διαβούλευση, είτε οι ε, κοινωνικοί εταίροι θα ε, συμφωνήσουν μεταξύ τους, είτε εμείς θα νομοθετήσουμε. Τώρα, η οδηγία για την γρατή δήλωση ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, καλύψει εκατομμύρια ατόμων τα οποία μετακινούνται και εργάζονται διασυνοριακά. Θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να τους καλύψουμε με ποια κριτήρια στην οδηγία. Αυτό το συζητάμε με του κοινωνικού εταίρου. Επίση υπάρχει άλλο ένα θέμα, πέραν τη πληροφόρηση που πρέπει να δέχονται, ποια είναι τα ελάχιστα δικαιώματά του που θα μείωναν την επισφάλεια. Έχουμε δει ποιε είναι οι πρακτικέ τι οποίε υφίστανται και θέλουμε να μειώσουμε την ε, επισφάλεια διατηρώντας την ευελιξία στην αγορά εργασίας. η, εργασία η Κομισιόν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και θα υποβάλει ένα νομοθετικό κείμενο στο τέλος του χρόνου περίπου. Αυτά και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους της Γενικής Διάθεσης Ανθρωπίνων Πόρων. Κύριε Καρλίνη και μετά ο κύριος Ροκ. Ε, η παρέμβασή μου θα επικεντρωθεί κυρίως ε, στην ε, πτυχή που αφορά τους ε, συμβασιούχους ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τμήματάρχης του τμήματος υπεύθυνου για τις προσλήψεις τους. Όσον αφορά τους συμβασιούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι δημιουργήθηκαν με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του 2004. Πριν από το 2004 υπήρχαν οι ε, επικουρικοί υπάλληλοι και πρέπει να πούμε ότι από το 2004 μέχρι σήμερα το ποσοστό των ε, εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου έχει μείνει το ίδιο. Δεν έχει υπάρξει αύξηση λοιπόν του αριθμού των συμβασιούχων σε σχέση πριν από 15 χρόνια. Ο αριθμός του σήμερα αυτών που έχουν συμβάσεων ε, ορισμένου χρόνου είναι περίπου 10% του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατ' ουσίαν ανταποκρίνονται ε, σε κάποια καθήκοντα τα οποία αφορούν ε, πολύ συγκεκριμένε ε, δραστηριότητες και δεν είναι ε, καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων. Δεν μπορούν να ασκήσουν κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα, δεν έχουν συγκεκριμένε αρμοδιότητες και υπάρχει μια διαδικασία επιλογής που είναι διαφορετική από την επιλογή των μονίμων υπαλλήλων. Εμεί θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η συμβασιούχοι ε, ου μόνον είναι απαραίτητοι για τη ζωή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και πολύ σωστή ρύθμιση. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ε, και που ανακύπτει από καιρού καιρών είναι το γεγονό ότι οι ε, ε, συμβασιούχοι δεν ξέρουν τι θα γίνει με τη σύμβασή του. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλή τι θα γίνει. Η μέγιστη διάρκεια που ήταν μέχρι τριών ετών μέχρι το 2014 αυξήθηκε με την τελευταία αναθέτηση αναθεώρηση του ε, κανονισμού των ε, υπαλλήλων και έγινε έξι χρόνια ε, μέγιστο. Ε, ένας ε, συμβασιούχος λοιπόν ο οποίος προσλαμβάνεται σήμερα ξέρει επακριβώς ότι μπορεί να εργαστεί το πολύ μέχρι 6 χρόνια ακριβώς για να αποφυγεί οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια διευκρινίζεται στην αρχή της σύμβασης και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά τις συμβάσεις είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει ένα κανόνα βάσει του οποίου συσσωρευμένες ε, ε, προσλήψεις ε, ε, αφορούν και κάποιους πυρογνώμονες αποσπασμένους εργαζομένους. Αυτοί δηλαδή που έχουν αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πάνω από 7 χρόνια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν χρησιμεύουν ε, για να διευκρινίζουν ευθύ εξ αρχής ε, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου και να διασφαλίζουν ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει και σεβασμό και ισορροπημένη διαχείριση των συμβασιούχων αυτών και προ το συμφέρον τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπής αλλά και για τους ίδιους εργαζομένους. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο ανέφερε ο κύριος Άσπρουκ ε, αφορά τους διαγωνισμούς για τους ε, συμβασιούχους εργαζομένους, τη δυνατότητα δηλαδή να μονιμοποιηθούν. Καταρχάς ε, θα ήθελα να διορθώσω ένα στοιχείο από αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Άσπρουκ που είπε ότι υπάρχουν μερικοί συμβασιούχοι που έγιναν ε, μόνιμοι υπάλληλοι. Από τον τελευταίο διαγωνισμό του 2016 έχουμε 30 υπαλλήλου. Και υπάρχουν άλλοι τόσοι που ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσλάβουμε ε, σύντομα. Όπως προφανώς γνωρίζετε υπάρχει περιορισμός ε, για την πρόσληψη των συμβασιούχων που καθορίζεται ε, από το καταστατικό και έχουν και λόγο ύπαρξη, διότι ένα από του λόγου για του οποίου. καθορίζονται είναι ότι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αντανακλά ε, τον ε, απαιτούμενο αριθμό. Δηλαδή, ε, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γεωγραφική ισορροπία των συμβασιούχων, το να προσλαμβάνουμε αδιακρίτως συμβασιούχους για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς διαγωνισμούς, θα μπορούσε να διαταράξει την γεωγραφική ισορροπία, την οποία προσέχουμε ιδιαιτέρως. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, διότι... Ούτως ή άλλως ε, αυτέ οι συνεδριάσει αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για να παρουσιάσουμε όχι μόνο τις νομοθετικές πτυχές αλλά και τις πτυχές τη πολιτικές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ σε μία πρόσφατη αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τους ε, συμβασιούχους ε, δεσμεύτηκε να γίνει ένας δεύτερος ανοιχτός διαγωνισμός για τους συμβασιούχους μέχρι το τέλος ε, της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι το τέλος του 2019 δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και που το χρονοδιάγραμμα. Ο επόμενος ομιλητής. Ο κ. Ροκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω ορισμένα από τα επιχειρήματα των αναφερομένων για να σας διευκρινίσω ε, ε, σε σχέση με την οδηγία και την αναφορά στο, στην απόφαση ότι στην απόφαση του δικαστηρίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει πολλές φορές κλπ. Το θέμα ήταν το κατά πόσον μια οδηγία εφαρμοζόταν στους συμβασιούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο, γιατί η οδηγία 9970 αλλά και γενικότερα οι οδηγίες ε, δεν απευθύνονται στις, ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο, το καταστατικό προβλέπει ένα μηχανισμό που, σύμφωνα με τον οποίο οι μόνες οδηγίες που εφαρμόζονται τα όργανα είναι αυτές που έχουν σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των αζωμένων στον χώρο εργασία. Ε, το δικαστήριο του Άνστρακ ε, αποφάσισε ότι το γεγονός πως ε, δεν λήφθη υπόψη η προστασία του, των διακοπών, των ημερών εργασίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία και πράγματι εκεί χάσαμε αλλά αυτό, αυτή η απόφαση αφορούσε ε, την άμεση εφαρμογή μια οδηγία στους υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η εξαίρεση. Να σας υπενθυμίσω ε, και το εξή Οι, οι αναφέροντες ε, κατηγορούν κατά κάποιο τρόπο τον νομοθέτη ότι δεν σεβάστηκε την οδηγία 9970 και μέσω του κανόνα των έξι ετών δεν την σέβεται. Όμως, ακόμα και αν δεν εφαρμόζεται κατευθείαν διότι πρόκειται για μια οδηγία πλαίσιο που δεν είναι άμεσα μεταφερόμενη στις, στα όργανα η, ο κανόνας των έξι ετών πράγματι γίνεται σέβεται την οδηγία και το 2004 και το 2013 ακριβώς σέβεται την οδηγία ο κανόνας αυτός σέβεται την οδηγία είναι η, παρα, η παράγραφος 5 του παραρτήματος προβλέπει μια, ένα μέγιστο όριο ε, διάρκειας ε, των ε, συμβάσεων, των συμβασιούχων. Ε, ο, το καταστατικό του 2013 ήταν σαφές. Αυτό που έκανε ήταν να πει ότι έχουμε τρία χρόνια μέγιστη διάρκεια που αν, αυτό, αν δεν ικανοποιούν τις ανάγκες ε, θα μπορούσαν αυτά τα τρία χρόνια να αυξηθούν σε έξι χρόνια. Οπότε από νομικής ε, πλευράς προφανώς και συμβαδίζουμε με την οδηγία. Δεύτερον, το δικαστήριο ποτέ δεν αμφισβήτησε ούτε το καταστατικό, τον εσωτερικό ανοισμό, ούτε ε, και την δυνατότητα χρήσης ε, τέτοιου είδους συμβάσεων περιορισμένου χρόνου. δύο αποφάσεις τα δύο τελευταία χρόνια, η μία από αυτές πολύ πρόσφατη, ε, απέρριψαν τις ε, προσφυγές ε, συνδικάτων, το U4U και το US, και το δικαστήριο διατήρησε τον ιστορικό στη μορφή που είχε το 2013. Μετά, άλλες αποφάσεις, Μαρία Ελένα Λόπες κλπ, διατήρησαν και πάλι τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου όπως έχουν. Οπότε όχι μόνο ο νομοθέτης δεν έχει παραβεί νομοθεσία, είναι αντιθέτως ε, έχει μεριμνήσει για το, την, ε, να γίνει σεβαστή η νομοθεσία και ο εσωτερικός κανονισμός. Τέλος, να προσθέσω αυτό που είπε ο Ρομπέρτο Καρλίν το εξή. Στον ε, περιορισμό των εξιετών και στον περιορισμό Τη πρόσβασης των συμβασιούχων σε εσωτερικού διαγωνισμούς, ε, δεν, πίσω από αυτόν τον περιορισμό δεν κρύβεται μόνο η προστασία τη γεωγραφικής κατανομής, αλλά και η προστασία του κινδύνου του νεποτισμού. Γιατί ε, η επιλογή των ε, συμβασιούχων γίνεται όχι με βάση διαγωνισμό, αλλά με βάση αυτού που βρίσκονται πιο κοντά στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Λουξεμβούργο, Ίσπρα, Βρυξέλλε. Και θέλουμε να μειώσουμε την περίπτωση νεποτισμού στην, στην μονιμοποίησή του. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Οκτώ ήταν οι ομιλητέ, Μεγάλη πρόκληση. Θέλω να αφήσω τη δυνατότητα και το χρόνο στους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ όμως να είστε πολύ πολύ σύντομοι. Εντουάρ και κυρία Εύη. Μια συνολική παρατήρηση. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή την ακρίβεια του κύριου Ροκ. Ήταν πραγματικά πολύ ακριβής. Αλλά ε, είμαι και ευρωβουλευτής και νομοθέτης. Ε, οπότε μας θέτεται ενώπιον των ευθυνών μας όταν ο νομοθέτης ψηφίζει ένα κείμενο, υπάρχει το κείμενο και το πνεύμα του κειμένου, του νόμου. Εμείς πολλές φορές ε, νομίζουμε ότι κάνουμε το σωστό, αλλά τελικά το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Παρακαλώ πολύ να μου εξηγηθεί κάποια στιγμή ε, το εξής. Οι ε, συμβασιούχοι καλύπτουν ανάγκες προσωρινής αύξησης του φόρτου εργασίας ή ασθένειες κλπ. Ε, ε, ε, το πρόβλημα είναι, θέλω να μου εξηγήσω το Αν οι ανάγκες είναι μόνιμες, που για ποιο λόγο τα συμβόλαια αυτά, οι συμβάσεις αυτές είναι προσωρινές και για την ίδια, για την ίδια θέση, μετά το τέλος των 6 ετών, της περίοδου των 6 ετών, προσλαμβάνεται κάποιος άλλος για άλλα 3 ή 6 χρόνια. Άρα λοιπόν η, η θέση αυτή είναι απαραίτητη και μόνιμη, ανεξάρτητα το αν καλύπτεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα από τον Α ή το Β. Αυτό δεν μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Δεν είναι σωστό αυτό. Οπότε, ε, ίσως πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία, έτσι ώστε το πνεύμα του νόμου να καταγραφεί και στο γράμμα. Thanks very much, um, Ναι, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στα όσα ακούστηκαν ε, για τις διαδικασίες επί παραβάση. Μάλλον, ε, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωση της Ιταλίας. Πώς είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχει ανάγκη να περιμένουμε για να γίνει αξιολόγηση όταν η πρώτη διαδικασία επί παραβάση ξεκίνησε το 2010 και άνοιξε λόγω των επισφαλών εργαζομένων στα σχολεία. Μετά έκλεισε επειδή υπήρχε νομοθεσία τη Ιταλία για τα καλά σχολεία που τελικά αποδείχθηκε καταστροφή για το σχολικό κλάδο. Ε, μετά ξεκίνησε μια άλλη διαδικασία που είναι ακόμα ανοιχτή, είναι εν εξελίξη και παρόλα αυτά η αμέλεια κατά την άποψή μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να διερευνήσει αποτελεσματικά ε, ε, παραβιάσεις κατά την άποψή μου κατάφορε τη οδηγία 9970, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφάρμοσε ούτε για την Ιταλία ούτε για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τις αρχές ε, οι οποίες έχουν εδρεωθεί πλέον στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επομένως κανένα, με κανένα τρόπο δεν κατάφερε να εγγυηθεί ότι θα εισαχθούν κατάλληλα αποτελεσματικά μέτρα στη κράτη-μέλη για να αποφευχθεί η κατάχρηση των συμβάσεων. Και να περάσω απευθεία στην ερώτηση, που πέραν από ερώτηση είναι μάλλον πρόταση, γιατί θα ήθελα ε, να αναφερθώ στους συναδέλφου όσον αφορά τον ευρωπαϊσμό. Και αυτό που μάθαμε ουσιαστικά από αυτή την ακρόαση ε, ε, είναι ε, ότι πρέπει να φτάσουμε στην Ολομέλεια με μια πολιτική εικόνα ενός θέματος, το οποίο έχουμε αμελήσει μέχρι τώρα και θα πρέπει εκ νέου μεθένους να μπει το θέμα αυτό στην επόμενη ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Ευχαριστώ. Ο Γιάρος Λαβαλέσα. Ευχαριστώ. Ποιες είναι οι συνέπειες για τους εργαζομένους, τι επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας όταν υπάρχουν διάφορες μορφές ε, άτυπης μορφής εργασίας και ποια ε, θα πρέπει να είναι οι πρώτες προτεραιότητες για τη δράση του ILO σε αυτή την περίπτωση ε, για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των βασικών αρχών, το δικαίωμα στην εργασία και άλλα δικαιώματα εργαζομένων σε μη ε, τυπικές μορφές ε, εργασίας. Τι προτεραιότητες θα πρέπει να υπάρχουν και πώς μπορούν ε, τα διεθνή εργασιακά πρότυπα να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις άτυπες μορφές εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι να υπάρχουν εάν υπάρχουν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, η κυρία Φορέντσα. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία την Επιτροπή αυτή. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά με ενδιέφερε ιδιαίτερα να παρέμβω για αυτό το θέμα, το οποίο παρακολουθώ όσο μπορώ και θεωρώ ότι εκπροσωπούμε, διότι και εγώ για 12 χρόνια ήμουνα επισφαλής εργαζόμενος του Πανεπιστημίου του Ιταλικού κράτους. Και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ όποιον την παρουσίαση. Θεωρώ ότι η παραβίαση της οδηγίας 9970 είναι προφανής ότι πολύ καλά κάνουν αυτοί που παρουσίασαν αυτή την αναφορά και την υποστηρίζουν να παρουσιάσουν και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ευθύνες ε, ε, της Ιταλικής Κυβέρνησης. Εύχομαι η διαδικασία επιπαραβάση όχι μόνο να ξεκινήσει, αλλά να ξεκινήσει πολύ γρήγορα, διότι στο μεταξύ οι συστηματικές παραβιάσεις ε, τείνουν να νομιμοποιηθούν. Το Jobs Act και το Buona Scuola, οι νομοθεσίες της Ιταλίας, ήταν ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μόνο στους ευρωβουλευτές μπορώ να δώσω το λόγο, λόγω του ε, σφιχτού χρονοδιαγράμματος. Μόνο 10 λεπτά έχουμε για τις απαντήσεις, το οποίο θα απαιτήσει και αυστηρή πειθαρχία από τους ομιλητές μας. Με αντίστροφη σειρά θα ξεκινήσουμε, διότι έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες ε, ερωτήσεις ε, απευθύνονταν ε, στους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ρωτήσω όμως, είναι δυνατόν μόνο ένας από εσάς να πάρει το λόγο από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. και αν ο κάθε ομιλητή μπορεί να περιοριστεί στο ένα λεπτό, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μου μαλώσει η πρόεδρο τη επιτροπή μα, διότι δεν θα φάω χρόνο από την ε, από τις δικές της τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τους συμβασιούχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν δύο στοιχεία κατ' ουσίαν. Το ένα αφορά ε, τις εξειδικευμένες ε, αλλαγές. αν δούμε ε, σήμερα τι ακριβώς γίνεται. Η πρώτη διεύθυνση που χρησιμοποιεί τους εργαζομένους ε, με ορισμένου χρόνου είναι η Γενική Διεύθυνση Έρευνες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, συχνά έχουν διδακτορικό ε, δίπλωμα και είναι ερευνητές. Και είναι απόλυτα προφανές ότι όταν πρόκειται για θέματα επιστημονικής φύσεως υπάρχει ανάγκη η οποία θα μπορούσε να είναι περιορισμένη χρονικά. Ε, το τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 5-6 χρόνια δεν θα είναι ακριβώ το ίδιο με σήμερα, με τι αλλαγές και τις συχνότητα των αλλαγών που βλέπουμε και τι κρίσει που έρχονται διαδοχικά η μία μετά την άλλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθησία. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε, και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο και το έθιξαν ε, κάποιοι παρουσιάσει του, ότι ενώ σε κάποια κράτη-μέλη οι διαγωνισμοί έχουν σταματήσει ή ε, δύσκολα μπορούν να γίνουν, όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπάρχει ο ΕΠΣΟ, ο οργανισμός ο οποίος διεξάγει διαγωνισμούς ετησίους και φυσικά οι συμβασιούχοι μπορούν να συμμετέχουν και σε αυτούς τους εξωτερικούς διαγωνισμούς. Ευχαριστώ κύριε Σκόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις ακούστηκαν από ευρωβουλευτές από την Ιταλία ε, σχετικά με το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διώκει περιπτώσεις στον Ιταλικό δημόσιο τομέα. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση και, η, και ο στόχος αυτών των διαδικασιών είναι η νομοθεσία των κρατών μελών να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Όπως σας είπα, μόλις ενημερωθήκαμε σχετικά με την Ιταλική νομοθεσία που τροποποιεί τις προϋποθέσεις για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα και για τους δικαστές. Τώρα πια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύσει να εξετάσει προσεκτικά την νομοθεσία αυτή και να διαπιστώσει εάν έτσι συμμορφώνεται η Ιταλική νομοθεσία με την ε, οδηγία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ε, εργαζόμαστε λοιπόν σκληρά πάνω στο θέμα αυτό. Η σχετική νομοθεσία ε, είναι του καλοκαιριού, λίγες εβδομάδες ηλικία έχει δηλαδή. Όσον αφορά το ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα ε, εργασιακά πρότυπα. Ε, θα ήθελα να επικροτήσω την ομιλία που ακούσαμε στην αρχή που περιείχε πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης. Επίσης υπάρχει έκθεση ε, της Επιτροπής την οποία πολύ ευχαριστώ θα διανύουμε εδώ στους συναδέλφους που παρουσιάζει την θέση της Επιτροπής σε σχέση με τις προκλήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ δίνω το λόγο στους άλλους ομιλητές. Παρακαλώ περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Ήμουνα κάπως πιο ε, επίοικης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι οι περισσότερες ερωτήσεις ε, απευθύνονται σε αυτούς. Ο κύριος Άσπροκ, πολύ σύντομα. Ε, ναι, όσον αφορά το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ε, μπορώ να σας πω ότι η Σύμβαση Υπαριθμών 98 επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη και από το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 50 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμορφώνεται καθόλου με τη σύμβαση αυτή. Ε, μάλλον θεωρεί ότι είναι υπεράνω, το οποίο μα δίνει μια ιδέα των σχέσεων ανάμεσα στη Γραφείο Εργασία, στον ILO και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γκαλεάνο. Πολύ σύντομα, μόνο μια σκέψη. Ο νόμος Μαντία για την μονιμοποίηση είναι από τις 25 Μαΐου του 2017. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω και τους χρόνους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά είμαστε στα τέλη Νοεμβρίου. Είναι δυνατόν ακόμα να μην μπορέσετε να εξετάσετε ε, το θέμα. Πέστε μου απλώς ε, τι χρονοδιαγράμματα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νόμιζα προχωράτε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ κύριος Δεμικέλε. Είναι πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει το κοινοβούλιο μόνο του. Ε, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 7 μέρες, την 7η ξεκουράστηκε βέβαια. Ο Ρουμάνος δικαστής Ντόντερ σε 6 μέρες επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη ε, προσφυγή για μην συμμόρφωση στην Οδηγία 99-70 Σε 7 ημέρες, εάν πιέσετε δεόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί όλες αυτές οι επισφαλείς καταστάσεις να οδηγήσουν σε μια ταχεία διαδικασία επιπαραβάση συνολικά και μια ταχεία λύση των προβλημάτων των ε, επισφαλών εργαζομένων στο δημοσιο όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you. Uh, Uh, Δεν υπάρχουν ερωτήσει για μένα νομίζω, αλλά έχω εγώ μια ερώτηση. Ποια είναι η συνέχεια που θα δοθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εδώ και πέρα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Επιτροπή είπε ότι για το, οι δύο αναφορές ε, του Βρετανίας και του Βελγίου ε, θα απαντηθούν εν καιρό ε, ξέρω ότι στείλατε ε, επιστολές στις εταιρείε. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε με τους αναφερόμενους τις απαντήσεις που θα λάβετε. Από την ε, πλευρά της Business Europe των εργοτών δεν υπήρχε κανείς εδώ νομίζω σήμερα. Ε. Οπότε τι συνέχεια θα δοθεί στις αναφορές. Πώς η σημερινή ακρόαση θα επηρεάσει την έκβαση. Ε, Δεν νομίζω μου τέθηκε καμία ερώτηση. Μπορείτε να περάσετε στο κλείσιμο. Θαύμα. Τελειώσαμε και λίγο πριν το χρόνο μας, ε, μας Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Από τη δική μου οπτική γωνία αυτές οι αναφορές είναι ανοιχτές και θα τις παρακολουθήσουμε εμείς ως ευρωβουλευτές από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Οπότε η συζήτηση θα συνεχιστεί και στο μέλλον προσπαθώντας να εντάξουμε σε αυτήν και τα σχόλια που είναι σήμερα και τις σημερινές παρεμβάσεις, τη γνώση που αποκτήσαμε κλπ. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε να ενσταλλάξουμε και όλα αυτά και στις υπόλοιπες εργασίες του Κοινοβουλίου, στις υπόλοιπες επιτροπές εξίσου όχι μόνο στην Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω ότι έχουμε αυτό τον ρόλο του διαμεσολαβητή έτσι ώστε όλα αυτά που γίνονται εδώ να εντάσσονται και στι υπόλοιπε εργασίε του Κοινοβουλίου. Το γεγονό ότι υιοθετήθηκε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, επισφαλή εργασία είναι δείγμα ότι οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν εν γέννη πως η αύξηση της ε, ε, επισφάλειας είναι κάτι αρνητικό για την κοινωνική Ευρώπη, για την κοινωνική συνοχή, για τον ε, κοινωνικό ιστό. Καθώς επίσης ε, αρνητική και για την οικονομία. Αν σκεφτώ τη δική μου πατρίδα, ε, που έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων μηδενικού χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ταυτόχρονα έχουμε και τα μεγαλύτερα κενά σε θέσεις εργασία υψηλών προσόντων. Ε, και αν δεν λοιπόν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, ασφάλειας στην εργασία, το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης κλπ, τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίξαμε σήμερα, ε, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά, υποσκάπτουμε την μακροβιότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέλος, να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχει μια διαβροτική τοξικότητα στο φαινόμενο αυτό, κάτι που θα έχει μακροπρόθεσμα πολιτικά αρνητικά αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Οπότε τα λόγια πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Χρειάζεται να περάσουμε στην ε, νομοθετική διάσταση του κοινωνικού πυλώνα. Νομίζω ότι πρώτη φορά καταφέρω να προεδρεύσω και να σεβαστούμε τους χρόνους μας. Δίνω ξανά το λόγο σε Σίλια. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις συνεισφορές. Δυστυχώς ε, δεν κατάφερα να είμαι μαζί σας το απόγευμα και να προεδρεύσω. Να υπογραμμίσω ότι το σημείο αφετηρίας ήταν πράγματι οι αναφορές ε, τις οποίες έχουμε λάβει και οι αναφορές αντικατοπτρίζουν τις ε, τελευταίες αλλαγές στον κόσμο της αγοράς εργασίας τις ε, τάσεις θα έλεγα, τις τάλ τάσεις. Τάσεις, καινούριες τάσεις οι οποίες φέρουν μαζί τους και προκλήσεις βέβαια. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι το να είναι κανείς επισφαλής εργαζόμενος είναι κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο, διότι η επισφάλεια στην εργασία επηρεάζει και την υπόλοιπη ζωή του εργαζόμενου. Οπότε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη καθώς επίσης και οι εργοδότες θα πρέπει να περιορίσουν στο μέτρο του δυνατού την έκθεση των εργαζομένων σε αυτό το φαινόμενο. Και κοινό μας στόχος θα πρέπει να είναι να προωθήσουμε τις αξιοπρεπείς ε, συνθήκες εργασίας, ε, την ισότητα, την αυτονομία, την ανεκρατησία των εργαζομένων. Και χαίρομαι που η Επιτροπή μας σήμερα αφιέρωσε πολύ χρόνο σε αυτό το φαινόμενο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το τμήμα πολιτικής, το αρμόδιο τμήμα πολιτικής, το οποίο πραγματικά μας παρουσίασε μια πολύ, πολύ ψηλής ποιότητος έκθεση. Θα είναι χρήσιμη αυτή η έκθεση όχι μόνο για τα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά και για όλο το όργανο και για άλλα όργανα και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και θεωρώ ως μικρό φως στην άκρη του τούνελ ότι έχουμε πλέον τον κοινωνικό πυλώνα. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι πια ένα απόμακρο όνειρο. Δεν είναι μια οπτασία. Είναι κάτι το πραγματικό, το απτό, στο οποίο, για το οποίο έχουμε αναλάβει δεσμεύσει. Α πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για ένα καινούριο ταξίδι, το οποίο μα περιμένει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά βέβαια. Ευχαριστηθείτε τα. Καλό σας βράδυ.